Good morning, dear colleagues, ladies and gentlemen. Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Good morning. Good morning to you all. Thank you for being here. Καλημέρα και πάλι. Καλώς ορίσατε. Of this Committee Inquiry on the electronic mass surveillance on EU. Ξεκινάμε τη σημερινή έρευνα ακρόαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών όσον αφορά τις μαζικές παρακολουθήσεις από την NSA. Θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά στη μερίσια διάταξη καταρχήν και να πω ότι σήμερα θα κάνουμε μια τρίτη ακρόαση ε, στο πλαίσιο της έρευνας για τις μαζικές ε, παρακολουθήσεις Ευρωπαίων πολιτών. Μέχρι στιγμής έχουμε μια ανταπόκριση και ενημέρωση, αλλά η σημερινή ακρόαση που είναι ιδιαίτερα εντατική θα περιλαμβάνει πέντε ε, συνεδρίες. Καταρχήν, ο συνάδελφος Μωράης Από το δεν τον είδα, δεν τον είδα. Ναι, ναι, βεβαίως, δεν σα είδα. Ε, ε, ίσως θα ήθελα να μας πει, να μας πει την ειδική οργάνωση της σημερινής ε, ε ημερήσιας διάταξης. Κλόντ, μπορείς να το σχολιάσεις λίγο. Ναι, ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω ένα-δυο παρατηρήσεις. Οι συνάδελφοι θέλουν να συνεδριάσουν, μάλλον, να, μάλλον ήρθαν σε μένα σε, ως εισηγητή για να τους ενημερώσω για τις διάφορες εξελίξεις καθώς θα συνεχιζόταν η έρευνα. Μάλιστα να πω ότι κάθομαι εδώ γιατί η γραμματεία δοκιμάζει διάφορες άλλες ρυθμίσεις για το που θα κάθονται οι σκιώδες και οι εισηγητές. Οπότε παρακαλώ λίγο υπομονή. Ε, ήθελα να σας ενημερώσω για το ποιος καλούμε και ποιοι δέχτηκαν τις προσκλήσεις μας σε αυτήν την ε, ακρόαση. Όπως έχουν τα πράγματα, έχει σταλεί ε, πρόσκληση στον Ρόμπερτ Γουάρντορ που είναι ο πρώτος γραμματέας και εν ενεργεία πρέσβης στην πρεσβεία των ΙΠΑ στην Ένωση, αλλά δεν λάβαμε επικύρωση ότι θα παραβρεθεί στη σημερινή μας ε, κρόαση. Ε, εστάλησαν και άλλες προσκλήσεις προς την Αμερικανική κυβέρνηση. Επίσης έχουμε καλέσει τους τον Ολλανδό Υπουργό Άιβο Όμπουσεν, καθώς και τον Ρόλαν Πλάστερ, πρώτος Υπουργό Δικαιοσύνη και ο δεύτερος Υπουργό Εσωτερικών, στην τρίτη συνεδρία για σήμερα, δεδομένου ότι η υπηρεσία SWIFT έχει έδρα στην Ολλανδία. Δυστυχώς και οι δύο υπουργοί ε, απέρριψαν την πρόσκλησή μας, ε, προτιμούν ε, τις ε, διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται ανάμεσα στην Επίτροπο Μάλστρομ και τον Υπουργό, ε, τον Γραμματέα Κόεν. Ενημέρωση για κάθε επαφή που είχαμε με την Αμερικανική κυβέρνηση. Και καθώς θα προχωρά αυτή η έρευνα και η εκρόση θα προσπαθήσω να σας ενημερώνω διαρκώς για το ποιος δέχεται και ποιος απορρίπτει τις προσκλήσεις μας. Ευχαριστώ. Κλοντ, ευχαριστώ. Υπάρχουν ε, αντιρρήσεις για την ατζέντα. Όχι. Εγκρίνεται τότε και περνάμε στην πρώτη από τις πέντε συνεδρίες που έχουμε προγραμματίσει. Θα κρατήσει μία ώρα και το πρώτο σημείο είναι οι αποκαλύψεις που είχαμε ότι Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσει στα νέα, υπήρξαν παρακολουθήσεις ε, και ε, στοιχείων από την βάση δεδομένων SWIFT από πλευράς της ε, NSA. Όπως ξέρετε, έχουμε γράψει την συμφωνία TFTP από, από το 2010 και εφεξής και επιτρέπεται η μεταφορά στοιχείων SWIFT μόνο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή της οικονομικής τρομοκρατίας. Η Europol έχει αναλάβει να επαληθεύει κατά πόσο τα αιτήματα των Αμερικανικών αρχών συμφωνούν με τους όρους ή όχι. Αυτός, αυτός ο όρος ήταν ένας από τους βασικούς ώστε να δεχτεί το Κοινοβούλιο αυτή τη συμφωνία ε, καταρχήν και έχουμε μαζί μας την Επίτροπο Μάλμστρομ που στις 12 Σεπτεμβρίου ε, στείλε επιστολή στον Υπουργό Κοένα, τον είπα, ζητώντας διευκρινήσεις. Ε, λάβαμε απάντηση στις 18 Σεπτεμβρίου. Το θέμα είναι προσυζήτηση στις 8 Οκτωβρίου. Αλλά σήμερα τους ή άλλως είμαστε πολύ ευτυχείς που καλωσορίζουμε ακόμη μια φορά ενώπιον της Επιτροπής Λίμπε την Επίτροπό μας, στρώμα και μετά θα έχουμε και τον ε, Διευθυντή της Europol, τον κύριο Winbright, και την κυρία Πέτρε από το SWIFT που θα μας ενημερώσουν για τα διακυβεύματα. Data Protection Supervisor. Έπειτα θα έχουμε τον Βέλγο αρμόδιο ε, ε, εποπτεία των στοιχείων, τον κύριο Ντεπόιτερε, αν το προφέρω καλά το όνομά του, πρέπει να είναι στην αίθουσα. Το Βρετανό μάλλον οι Βρετανικές ε, αρχές διερευνούν και την υπόθεση της παρακολούθησης από την NSA, μάλλον της ανάμειξης NSA στα συστήματα της βελγικής Belgacom. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην Επίτροπό μας για μια σύντομη ε, δήλωση όσον αφορά την, τα στοιχεία που παίρνει η από την βάση δεδομένων SWIFT και τις επιπτώσεις που θα έχει αυτός για τη συμφωνία μας. Και έπειτα θα έχουμε ερωταπαντήσει. Επειδή έχουμε όμως εντατική συνεδρία σήμερα με πέντε συνεδρίες, προτείνω όλοι όσοι θέλουν να πάρουν το λόγο και να συμβάλλουν στη συζήτηση να περιοριστούν στο δίλεπτο. έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για τους υπόλοιπους προσκεκλημένους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την Επίτροπο. Κυρία Μάλαστρο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω ορισμένα στοιχεία σε σχέση με την πιθανολογούμενη πρόσβαση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνική Ασφάλειας στα δεδομένα που υπόκειται στη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένων Πολιτειών. Και θα εστιάσω στα θέματα αυτά γιατί ξέρω ότι άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την αντικατασκοπία θα αντιμετωπιστούν αργότερα. Ανησυχώ πάρα πολύ για αυτές τις ε, ε ειδήσει, τους ισχυρισμού που δημοσιεύτηκαν στον τύπο. Η συμφωνία TFTP με τις ΗΠΑ έγινε ακριβώ για να αποφύγει τα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών να βρίσκονται χωρί διαφυλάξει και νομικέ διασφαλίσεις. Ο στόχο ήταν να υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας τα οποία μοιραζόμαστε με τι ΗΠΑ ότι τα αντιμετωπίζονται με τρόπο σύμμορφο με την προστασία των προσωπικών δικαιωμάτων. Η συμφωνία αυτή καλύπτει επίση οποιαδήποτε μετάδοση δεδομένων από τη βάση δεδομένων SWIFT από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας έχω παρουσιάσει λοιπόν και στο παρελθόν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προστασία αυτών των δεδομένων στη συζήτηση των προγραμμάτων 2011 και 2012 και οι υπηρεσίε μου προετοιμάζουν μια έκθεση για το TFTP και την αξία του εν ώψη των πρόσφατων ομοσεξελίξεων ανεβλήθη αυτό 4 <clears throat> Ιουλίου. Μετά από τις πρώτες εκθέσεις για την ύπαρξη ενός προγράμματος Παρακολούθηση από τι ΗΠΑ του πρίσμα. Εγώ έστειλα μια επιστολή στον ομόλογο μου στι ΗΠΑ ζητώντα πλήρη σαφήνεια για τα προγράμματα αυτά και τι επιπτώσει του για το TFTP και επίση για τη συμφωνία PNR. Παραλίλω. η ομάδα εργασία για την προστασία δεδομένων οι Ηνωμένε Πολιτείε Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να εξετάσει τι ακριβώ συμβαίνει με τι καταγγελόμενε αυτέ παραβιάσει. Και είναι, ακόμα εν εξέλιξη αυτή η έρευνα. Στι αρχές Σεπτεμβρίου ήρθα σε επαφή με τον David Cohen από τις ΗΠΑ, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και του ζήτησα περαιτέρω πληροφορίες για το τι ακριβώς θα προκύψει ως απάντηση των ΗΠΑ για όλα αυτά τα θέματα. Του απέστησα και μία επιστολή όπου ζήτησα να ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις επί τη βάση του άρθρου 19 της συμφωνίας μας. Αυτό είναι ένα επίσημο βήμα το οποίο πρέπει να γίνει όταν υπάρχουν διαμάχες μεταξύ των δύο συμβαλωμένων μερών στη συμφωνία TFTP. Κατά τη διάρκεια αυτών των ε, συζητήσεων θα προσπαθήσω να αποσπάσω πλήρες πληροφορίες και εξηγήσεις για να μπορέσουμε να διακριβώσουμε σε ποιο βαθμό η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας μπορεί να έχει σημειωθεί. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έδωσαν στην απάντησή του στην επιστολή μου κάποιε εξηγήσει. Σας έχω διαβιβάσει αυτή την επιστολή. Τίθενται βέβαια μια σειρά από προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν βάσει τις διαδικασίες του άρθρου 19 τη διαβούλευση. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένο από τι απαντήσει που έχουμε λάβει μέχρι στιγμή. Υπήρχε μια κατανόηση από την πλευρά των ΗΠΑ, αλλά δεν μα έχουν δοθεί πλήρε πληροφορίε για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ποια είναι η πραγματικότητα και να δούμε κατά πόσον έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσει τη Αμερικανική πλευρά ή όχι. Είναι το θέμα ύψη τη προτεραιότητα για μένα και τι υπηρεσίε μου να συνεχίσουμε τι διαβουλεύσει με τι ΗΠΑ. Θα συναντηθούμε πρόσωπο με πρόσωπο με του ομολόγου μα των ΗΠΑ πολύ σύντομα. Θα ήθελα να μου δώσετε ερωτήσεις που μπορώ να μεταφέρω στους Αμερικανούς ομολόγους μου και φυσικά εγώ θέλω να ομιλώ εξ ονόματος όλων των θεσμικών οργάνων. Συγκεκριμένα ερωτήματα θα ήθελα να έχω λοιπόν να μεταφέρω. Μία απόφαση λοιπόν είτε να διατηρήσουμε τη συμφωνία ή να προτείνουμε την αναστολή της είναι βέβαια ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Κατανοείτε ότι βέβαια τα δημοσιεύματα στη, στον τύπο μπορεί να δημιουργήσουν διαδικασία διαβούλευσης, μία αναστολή της συμφωνίας απαιτεί μία αντικειμενική αξιολόγηση και διαβουλευση. Χρειαζόμαστε πιο πολλές πληροφορίες, μεγαλύτερη σαφάνεια, σαφήνεια. Ελπίζω να τα αποκομίσω αυτά το ταχύτερο δυνατόν και θα σας κρατήσω απόλυτα ενήμερους για τις εξελίξεις αυτές και οποιαδήποτε πρόταση για το μέλλον της συμφωνίας TFTP θα πρέπει να συζητηθεί και μαζί σας. Κλείνω εδώ για να μπορώ να απαντήσω στα ερωτήματά σας κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ Επίτροπε Μάλστρομ για την δήλωση που κάνατε η οποία ήταν ε, πολύ γρήγορη, swift στα αγγλικά όπως λέμε και πολύ ακριβής ε, μέσα στο θέμα θα έλεγα. Έχουμε λοιπόν τώρα χρόνο για ερωτήσεις. Θα έλεγα πρώτα να μιλήσουν οι εισηγητές, μετά οι σκιώδεις και μετά οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Βέβαια δεν είναι μικρός ο κατάλογος των ομιλητών και για αυτή τη συνεδρία, για αυτή την ανταλλαγή απόψεων ε, και τις ερωταπαντήσεις με την Κομισιόν έχουμε χρόνο έως τις 10. Θα σας παρακαλέσω να περιοριστεί το καθένα στα τρία λεπτά. Αλλιώς, ε, ως συνήθως, θα μπλέξουμε. Κύριε Μωράης, πρώτος. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε. Σας ευχαριστώ επίσης πρόεδρε και εσάς κύριε Εύτρου που αφήσατε για μας τους βουλευτές χρόνο για ερωτήσει, είτε αυτό θέλουμε. Για την ενδεχόμενη αναστολή της συμφωνίας θα συζητήσω στο τέλος, αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφέρω σε αυτά τα οποία ε, είτε εν μέρη έχουν απαντηθεί είτε δεν έχουν απαντηθεί στην πρώτη σας επιστολή προς τον Υπουργό Κόεν, που θα πρέπει ενδεχομένως να τα ξαναθέσετε πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τις αποκαλύψεις που έχουν να κάνουν με τη δράση του Υπουργείου Οικονομικών των Πολιτειών. Το NSA που έχει πρόσβαση στα συγκεκριμένα γραφεία του Υπουργείου Οικονομικών, έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία του SWIFT ή κάπου αλλού. μήπως έχοντας άμεσα ή έμεσα πρόσβαση σε κάποια κέντρα ε, φύλαξη δεδομένων στην Ευρώπη γιατί δεν έχουμε κανένα στοιχείο πάνω σε αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε κατά πόσον ε, η NSA ή άλλες υπηρεσίες πληροφοριών ε, των ΗΠΑ είχαν πρόσβαση ε, στα στοιχεία SWIFT παραβιάζοντας διατάξεις της συμφωνίας TFTP και αν υπήρξε επίσης κάτι το οποίο μπορέσατε να εντοπίσετε και αν έχουν ληφθεί μέτρα. Στο άρθρο 12 της συμφωνίας SWIFT μιλά για την παρακολούθηση, για τον έλεγχο. Εκεί ζητείτε ξεκάθαρα να υποπτεύετε από, ανεξάρτητη, από ανεξάρτητο πρόσωπο ε, η εξέταση στοιχείων που έχουν να κάνουν με, με το SWIFT. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένας ανεξάρτητος επόπτης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης το άρθρο 8 του χάρτη για τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ξεκάθαρα ότι κανείς προστατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών, προστασία των δεδομένων μεταξύ αυτών, πρέπει να ελέγχεται από μια ανεξάρτητη αρχή. Τώρα, θα πρέπει η Κομισιόν να, να επανεξετάσει το μηχανισμό υποπτίας. Ίσως θα πρέπει να οριστεί ένας εξωτερικός EDPS. Δεν ξέρω αν και το Συμβούλιο συμφωνεί. Είστε έτοιμοι να κάνετε μια έκθεση για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του άρθρου 12. Παραδείγματο χάρη, αυτό ο ανεξάρτητο ε, εκπρόσωπο πόσε φορέ μπλοκάρισε ε, την πρόσβαση σε στοιχεία SWIFT ε, με βάση την τελευταία συμφωνία. Έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, έχουμε αποκτήσει νέες ευθύνες έκτοτε και ξέρουμε ποιο είναι πλέον ένα αποδεκτό επίπεδο προστασίας. Συμφωνείτε ότι το εν λόγω συμφάνα έχει πλέον καταστήσει σαφές ότι πρέπει να επανεξεταστεί και να επικαιροποιηθεί η συμφωνία αυτή ώστε να έχουν οι πολίτες την προστασία την οποία δικαιούνται. Και σε ό,τι αφορά τώρα την ενδεχόμενη αναστολή, ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει αρκετούς από εμάς, επειδή έχετε ξεκινήσει ε, κάποιες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας συμφωνία SWIFT. Πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το δεχόμενο αναστολή. σε Συμφωνείτε ότι πρέπει να ανασταλεί εφόσον δεν λάβατε επαρκή απαντήσεις από την Αμερικανική πλευρά και λόγω της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τώρα τον κύριο Άλβαρ, τον ε, εισηγητή μας ε, για το TFTP. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Σεσίλια, την Επίτροπο Μάλστρομ που βρίσκεται εδώ ιδίω γιατί σας ενδιαφέρει ο ρόλος ε, της NSA ε, είναι πάρα πολύ σημαντικός και πρέπει να γίνουν ε, σίγουρα κάποια τουλάχιστον στοιχειώδη πράγματα και κινήσατε και τις διαδικασίε δυνάμει του 19 της συμφωνίας τη FTP. Χαίρομαι γι' αυτό. Αν με επιτρέπετε θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις πάνω στη συμφωνία τη FTP. Συμφωνήσαμε περίπου τον, νομίζω τον Αύγουστο του 2010 η Κομισιόν να παρουσιάσει την 1η Αυγούστου του 2011 μια πρώτη πρόταση για το Αμερικανικό Σύστημα Εξαγωγής Δεδομένων και να μας αναφέρει για ένα αντίστοιχο σύστημα δυνάμει του άρθρο 11 της Συμφωνίας. θα μπορούσαμε να περιμένουμε σύντομα να έχουμε τέτοιες προτάσεις. Και έρχομαι στη συμφωνία. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας, τα δεδομένα τα οποία ζητούνται θα πρέπει να δίνονται όσο το δυνατόν πιο περιοριστικά. Και η Κομισιόν λέει ότι το Υπουργείο των ΗΠΑ δεν θα έχει ποτέ πρόσβαση σε ένα ευρύτερο σε τα ε, ζητούμενων δεδομένων. Εάν όχι, τότε γιατί τα διατηρούν αυτά τα δεδομένα. Τώρα έρχομαι στο άρθρο 16 που λέει ότι υπάρχει δικαίωμα επανόρθωσης για τα, πρόσπα, τα οποία, ε, των οποίων είναι τα δεδομένα που, στα οποία είχε πρόσβαση η NSA. Αυτή λοιπόν η επανόρθωση τεχνικά δεν ήταν εφικτή με αυστηρή τεχνική έννοια και πιστεύω ότι και αυτό μας δημιουργεί ανησυχίες. Το άρθρο 6 λέει επίσης ότι τα δεδομένα διαγράφονται το αργότερο 5 έτη από την παραλαβή τους ε, αλλά τα δεδομένα τα οποία τα έλαβαν ε, από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 7 δεν διαγράφηκαν μέχρι τα τέλη του 2012, άρα αυτό είναι ένα θέμα ακόμη. Για το άρθρο 12 τώρα συμφωνώ ε, με αυτό που είπε ο συνάδελφος Κλόντ Μωράης. Το ερώτημα που σας έθεσε και για να μην μακρηγορώ, επειδή περνάει ο χρόνος μου, θέλω και εγώ να συμφωνήσω και να στηρίξω τον Κλόντ Μωράης ε, στο θέμα της αναστολής, διότι το Κοινοβούλιο δεν μπορώ βέβαια εγώ να εκπροσωπήσω όλο το κοινοβούλιο εδώ. Προσωπικά όμως θα ήμουν υπέρ του να έχουμε τουλάχιστον ε, την αναστολή ως μια επιλογή, να συζητήσουμε το ενδεχόμενο της αναστολής αυτής της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και επίσης να ξεκαθαρίσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι, οι καζόμενες παραβιάσεις Έστω η αμφιβολία που υπάρχει ενδεχομένω ε, να είναι αληθινό αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει σε τίποτα άλλο από την αναστολή τη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Α ακούσουμε του κοιόδης εισηγητές και θα επανέλθουμε στην κυρία Επίτροπο και θα υπάρχει και λίγο περιθώριο να λάβουν το λόγο και τα υπόλοιπα μέλη. Ο κύριος Φως από το ΕΛΚ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Έχω ερωτήματα τα οποία είναι παρόμοια με αυτά τα οποία ανέφερε η Διοκλώτη Μωράη και ο Αλεξάνδρ Άλβαρος. Κατα... Καταρχήν, έχετε στοιχεία σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν αναφερθεί στις ε, εφημερίδες ότι η NSA έχει ένα τρόπο να παίρνει πληροφορίες κατευθείαν από το SWIFT ότι έχει κάποιο ε, κάποια προγράμματα ή κάποιους δούριους ύπους αυτού του είδους. Δεύτερον, έχετε κάποια στοιχεία που να αναφέρουν ότι η NSA ε, δεν πήρε μονάχα στοιχεία από το SWIFT, αλλά συνέχισε να παίρνει αυτά τα στοιχεία μέχρι και τη στιγμή που έγινε συμφωνία TFTP. Ποια είναι λοιπόν τα κομμάτια πληροφοριών που έχει πάρει η NSA πριν γίνει η συμφωνία και ποια είναι αυτά που είναι μετά τη συμφωνία. Και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και κάποιος πρέπει να το κάνει. Ή θα το κάνουμε εμείς ή θα το κάνουν οι Αμερικανοί. Από ό,τι κατάλαβα εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε και επομένως έχει επαφιεθεί αυτό στους Αμερικανούς. Η δική μου τώρα εντύπωση είναι, είναι ότι έχουμε δύο συνέχειες που θα πρέπει να δώσουμε. Καταρχήν, επί τη βάση της συμφωνίας που έχουμε κάνει για το SWIFT και με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την καταπολέμηση της ε, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες και έχουμε τώρα μια διαδικασία η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μη νόμιμη, ως ε, παράνομη. Δεν ξέρω λοιπόν αν πρέπει εμείς να καταγγείλουμε από τη μία πλευρά τη συμφωνία, αλλά να αφήσουμε την διαδικασία παράνομης συλλογής δεδομένων να την αφήσουμε να συνεχίζεται ή αν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα δύο με, με ένα συνεκτικό τρόπο. Intveld. Σας ευχαριστώ. Εγώ είμαι λίγο πιο πολιτική στα ερωτήματά μου. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι για τη στεναρότητα που έχει πάρει η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τον έναντι των ΗΠΑ. Οι απαντήσει που μας έχουν δώσει οι Αμερικανοί δεν μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικέ. Αν δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τη συμφωνία TFTP, ήταν αμφιλεγόμενη αυτή η συμφωνία από την αρχή. Η νομική της βάση είναι επίμαχη και αμφιλεγόμενη, για να το πω επί οίκος. Η δική μου πολιτική ομάδα έδωσε την έγκρισή της σε αυτή τη συμφωνία με τη λογική ότι η Κομισιόν θα έδινε, θα έκανε κάποιες προτάσεις για ένα σύστημα ε, για την ανάκτηση δεδομένων. Αλλά αυτό το σύστημα δεν υπάρχει. Αυτή η πρόταση της Κομισιόν δεν υπήρξε. Επομένως η προϋπόθεση για την έγκρισή μου δεν υπάρχει πια. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες για τον τρόπο που έχει εφαρμοστεί αυτό το σύστημα. Πολύ σημαντικές εκθέσεις θεωρούνται εμπιστευτικέ και τώρα υπάρχουν οι καταγγελίες ότι μπορεί η NSA <clears throat> να έχει άμεση πρόσβαση στους διακομιστές του SWIFT και επίσης να έχει χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για στόχους που δεν έχουν καμιά σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και έχουμε στοιχεία ότι το κάνουμε αυτό τουλάχιστον από το γεγονός ότι δεν το αρνούνται ήδη. Δεν ξέρουμε το κάνανε, αλλά η απάντησή τους είναι ότι εμείς επιφυλασσόμεθα στον εαυτό μας το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία. Είτε το έχουν κάνει μέχρι τώρα είτε όχι. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία λοιπόν γιατί επιφυλάσσουν στον εαυτό τους το δικαίωμα να κάνουν χρήση αυτών των δεδομένων. Κατά τη δική μου άποψη λοιπόν αυτή η συμφωνία είναι νεκρή και πεθαμένη. Έχει μονομερός καταγγελθεί στην πράξη. Εφόσον οι Αμερικανοί θεωρούν ότι δεν χρειάζεται μια συμφωνία για να ανακτούν τα στοιχεία και μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία για ό,τι σκοπό θέλουν, τότε αυτή η συμφωνία είναι πλήρως άκυρη και χωρίς καμία ισχύ. Εφόσον η επιστολή τους <clears throat> λέει ότι σέβονται μεν τη συμφωνία TFTP αλλά πίσω από τη βιτρίνα κάνουν ό,τι θέλουν, θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν αν είναι έτοιμη να ζητήσει την αναστολή αυτής της συμφωνίας ή καλύτερα σύμφωνα με τον κύριο Αλβάρο την απόλυτη καταγγελία και την ακύρωση αυτής της συμφωνίας. Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι το Κοινοβούλιο βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας έχει την ε, εξουσία να εγκρίνει διεθνείς συμφωνίες. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένα είδος <clears throat> επιταγής σε λευκό η του Κοινοβουλίου. Από τη στιγμή που έχουμε δεχτεί μια συμφωνία, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν είναι μια σημαντική δοκιμασία για τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν δεν έχουμε κανένα τρόπο να επέμβουμε σε τέτοιες συμφωνίες, εγώ θα είμαι ιδιαίτερα δεστακτική να προσυπογράψω οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία στο μέλλον. Είναι και ένα πολιτικό θέμα λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλμπρεχτ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ δεν θέλω επαναλάβω τα όσα ήδη υπόθηκαν. Ε, είναι σημαντική η ανταλλαγή αυτή απόψεων και θέλω να προσθέσω το θέμα Εάν δεν σκέφτεσαι αναστολή της συμφωνίας άμεσα, δέχεστε ότι υπάρχει πιθανή παραβίαση της συμφωνίας FTP, ωστόσο και θα κάνετε διαδικασίες κατά παράβαση κατά των ε, κρατών μελών που δεν πληρούν τους κανόνες για τα κυβερνο... εγκλήματα παραβίαση στα συστήματα από την NSA. Μπας περιπτώσει, τι, τι δράση θα αναλάβατε για την προστασία των συστημάτων ε, ε, πληροφοριών Τη Ευρωπαϊκή Ένωση που παραβιάζεται από την NSA ε, άλλες ε, ε, ομάδε κατασκοπίας όπως τη της πράγμα που είναι μέσα στι αρμοδιότητές σας φυσικά Σα ευχαριστώ η κυρία Έρνστ Το εξή ερώτημα θέλω να σα θέσω θα ήθελα να ξέρω από εσά, κυρία Μάλστον το εξή. αν υπήρξε κάποια ένδειξη, κάποια, κάποιος τρόπος να καταλαβαίνουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν παραδεχτεί έσω την ελάχιστη παραβίαση ή την έλλειψη πλήρους συμμόρφωσης με τη συνθήκη αυτή. Υπάρχει κάποια ένδειξη ότι το έχουν δεχτεί αυτό. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι Εσείς έχετε τώρα τα έγγραφα αυτά στη διαθέσή σας που χρειάζεται, κάντε τις απαραίτητες επαφές. Πώς είσαστε εσείς ως Επίτροπος σε θέση να καταλάβετε τι ακριβώς έχει γίνει. Έχετε δυνατότητα λοιπόν να έχετε όλη αυτή την τεκμηρίωση που αφορά αυτά τα προβλήματα και να μπορέσετε εσείς να είστε πεπισμένοι και να έχετε μια εμπεριστατωμένη γνώμη για το σε ποιο βαθμό έχουν παραβιαστεί οι διατάξεις της συνθήκης. Τρίτον, πώς γίνεται η προστασία <clears throat> των στοιχείων του SWIFT από διαβίβαση σε τρίτους. Πώς λειτουργεί στην πράξη αυτό το πράγμα και ποιος ελέγχει την ασφάλεια των δεδομένων μέσα στη συμφωνία SWIFT. Υπάρχει μια τέτοια επαλήθευση ασφάλειας και ποιος την κάνει. Άλλα αυτά τα ερώτηματα λοιπόν που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια για την μετάδοση στοιχείων του SWIFT μου είναι πολύ ενδιαφέροντα. εμένα. Επίσης, είναι σαφές ότι όπως είπε και η Σόφη Φανέλτ, η συμφωνία SWIFT δεν έχει κανένα νόημα γιατί όπως είναι φανερό οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται καν μια τέτοια συμφωνία για να αποσπούν δεδομένα. Και εγώ υποστηρίζω την καταγγελία αυτής της συμφωνίας. Και είναι προφανές για μένα ότι υπήρξε κατάχρηση αυτής της ε, συμφωνίας. Συνεχίζω τώρα εκεί που σταμάτησε η Σοφή. Πώς θα πρέπει να δράσουμε για να καταγγείλουμε αυτή τη συμφωνία. Τι προβλέπετε για να καταγγελθεί αυτή η συμφωνία. Τι θα έπρεπε να γίνει. Ποια είναι τα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να καταλήξουμε σε μια καταγγελία της συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, είναι σαφές ότι πολλά ε, από όσα ακούστηκαν συγκλίνουν μεταξύ τους. Βλέπουμε ότι αφισβητείται πολύ σοβαρά η συνέχιση ε, της ισχύωσης της συμφωνίας FTP. Πρώτα απ' όλα το Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσει αναστολή, να καταγγείλει ακόμη και την ίδια την συμφωνία, άρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Είμαι βέβαιος ότι θα μας ε, δώσετε μια πρώτη απάντηση και κάποια πρώτα στοιχεία με βάση την ανταλλαγή ε, και τις συνομιλίες που είχατε με τις αρχές ε, των ΗΠΑ και θα δώσω μετά το λόγο στους υπόλοιπους βουλευτές. επίτροπους. ευχαριστώ πολύ ε, που μου δίνετε το λόγο. Φυσικά και είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, εξού και βρισκόμαστε σήμερα εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ. Μπορούμε να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων Είμαι βέβαια ότι θα ακολουθήσουν και πολλές άλλες. Για να δούμε ε, το ιστορικό. Διαπραγματευτήκαμε με μια συμφωνία με τους Αμερικανούς για να έχουμε με, με αυτούς συνεργασία, για να μπορούμε να εντοπίζουμε ε, τους διάφορους χρηματοδότησης των ε, τρομοκρατών. Σοφ Ιντφελτ είπε ότι ήταν μια επίμαχη συμφωνία. Αλλά το Κοινοβούλιο τη δέχθηκε. Υπήρξε μάλιστα μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα, στη συμφωνία αυτή είχαμε σαφεί ασφαλιστικέ δικλείδε ε, για το στόχο, για το ποιο έχει πρόσβαση προστασία δεδομένων, πώ θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα και ούτω καθεξής. Ε, και θεωρήσαμε ότι υπάρχει επαρκή προστασία, εξού και συμφωνήσαμε. Έγιναν δύο αναθεωρήσεις, τις έχουμε συζητήσει και με εσά. Σε αυτές τις αναθεωρήσεις ε, φάνηκε υπήρχαν κάποιες αρχικές προκλήσεις που πρέπει να βελτιώσουμε, αλλά δεν ε, διαπιστώθηκε κάποιο ομίζον πρόβλημα ή κάποια παραβίαση της συμφωνίας. Ε, και επίσης έχουμε και ε, συνεργασία με την άλλη όχθη του Ατλαντικού για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα της εποπτείας και θα ολοκληρωθεί η έκθεση την οποία είχατε ζητήσει να γίνει με θέμα την προστάμενη αξία αυτής της συμφωνίας. Έχει γίνει ουσιαστικά αυτή η δουλειά, αλλά με τη συμφωνία αυτή ε, και τις συζητήσεις που έχουμε τώρα έχει μπει λίγο στο ψυγείο. Υπήρξαν πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες στον τύπο, πάρα πολύ ε, σοβαρές, δεν ξέρουμε κατά πόσο αληθεύουν ή όχι, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρές ε, ώστε να θέσουν πολύ σημαντικές ερωτήσεις εμείς να τους θέσουμε στους Αμερικανούς. Το κάναμε εμείς, το κάνετε κι εσείς και εγώ ε, με τηλεφωνική επικοινωνία αλλά και με αλληλογραφία τις ΕΡΣ αυτές τις ερωτήσεις. Και αν οι καταγγελίες αυτές αληθεύουν, σίγουρα συνιστούν παραβίαση της συμφωνίας. Και η παραβίαση της συμφωνίας φυσικά και μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή αυτή. Γι' αυτό το λόγο με βάση τη συμφωνία κιόλα ε, λέμε ότι ε, οποιαδήποτε αναστολή θα πρέπει να γίνει αφού προηγηθούν διαβουλεύσεις. Ζητήσαμε την έναρξη διαβουλεύσεων, οι οποίε θα ξεκινήσουν πάρα πολύ σύντομα. Έγινε μια ανταλλαγή αλλογραφία, σας ε, κοινοποίησα την επιστολή την οποία έλαβα εγώ, δεν νομίζω ότι απαντά τα ερωτήματα. Και δεν έχω λάβει Καμία άλλη προφορική ή γραπτή απάντηση. Κανένα είδο. κανένα υλικό δεν έχω λάβει. Και φυσικά και εμένα παραμένουν πάρα πολλέ απορίε μετά από αυτή την επιστολή. Εσεί είπατε ότι ε, θα πρέπει να δούμε ε, όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρονται στον τύπο και ένα-ένα να τα δούμε αν αληθεύουν ή ευσταθούν και πολλά άλλα θέματα. Όλα αυτά, όλα αυτά είναι επιτάπτωση και θα τα συζητήσουμε. Τώρα μπορούμε να κρίνουμε για το κατά πόσο υπήρξε έχει παραβίαση τη συμφωνία. είναι μια διεθνή συμφωνία, πρέπει να γίνουν κάποια συγκεκριμένα βήματα και μετά να καταλήξουμε. Και αν καταλήξουμε στο ότι ναι υπήρξε παραβίαση της τότε η Κομισιόν θα συζητήσει εσωτερικά το θέμα αυτό, ε, το Σώμα των Επιτρόπων ε, θα ε, αποφανθεί και αν αποφασίσουμε για αναστολή, αυτό θα αποφασιστεί από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Δεν έχουμε φτάσει εκεί όμω ακόμη, προηγούνται πολλά ακόμη να γίνουν, πολλέ απαντήσει να πάρουμε μέχρι τότε και να είστε βέβαια θα σα στηρώ πλήρως για όλα τα βήματα. Σε ό,τι αφορά τα ερωτήματά σα, δεν μπορώ να σα δώσω απαντήσει. Δεν τι γνωρίζω τι απαντήσει. Απλά θα τα εξετάσω όλα αυτά. Να πω στον κύριο Άλβαρο ότι ναι, αυτή η έκθεση για τι δυνατότητε εξαγωγή δεδομένων επί ευρωπαϊκού εδάφου. Ναι, πράγματι υπάρχει και υπό το φως των όσων ε, έγιναν. Έχει μπει λίγο, επαναλαμβάνω, το έχουμε βάλει λίγο ε, κατά μέρο ε, στο ψυγείο, θέλετε. Αλλά θέλαμε πρώτα να μελετήσουμε όλα τα στοιχεία και μετά να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Καταλαβαίνω, πρόεδρο, ότι δεν ε, είναι ικανοποιημένοι οι βουλευτές με τις απαντήσεις που δίνω, απλά μπορώ να σας δώσω απαντήσεις μόνο για όσα γνωρίζω. Ευχαριστώ και συνεχίζουμε με τους ε, υπόλοιπους. Έχουμε μακρύ καταλογό, οπότε παρακαλώ έχετε στο νου το χρόνο, γιατί πρέπει να ακούσουμε τον κύριο Ντεμποκαλίρ από την Belgacom και τον κύριο ε, το διευθυντή της Europol. Δύο λεπτά έκαστος ο κύριος Πίρκερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια εναρκτήρια παρατήρηση για μας ήταν σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα θέματα της τρομοκρατίας. Γι' αυτό μας φάνηκε απόλυτα λογικό να έχουμε συνεργασία με ένα σημαντικό εταίρο όπως οι Αμερικανοί. Και γι' αυτό έχουμε εξασφαλίσει και την ανταλλαγή πληροφοριών προς το στόχο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει ότι δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσει την απόλυτη ασφάλεια των ε, πληροφοριών τους και επίσης ξέρουμε ότι γίνεται κατασκοπία για στοιχεία τα οποία έχουν οικονομικό ενδιαφέρον για την οικονομική δραστηριότητα της Ευρώπης. Εδώ θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν αν θεωρεί ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας υπηρεσίας αντικατασκοπίας η οποία θα μπορεί να αποτρέπει την ε, ε, απόκτηση στοιχείων που έχουν να κάνουν με οικονομική δραστηριότητα και άλλα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι κάπου η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου έχει τονίσει την ανάγκη να υπάρξει μια συνεργασία στην αντικατασκοπία μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει όμως κάποια πρόταση από την πλευρά της Κομισιόν για ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό αντικατασκοπίας. Δεύτερον, έχει καταγγελθεί ότι έχουν ε, χρησιμοποιηθεί παράνομα. Έχουν ναι, αποσπαστεί στοιχεία από το SWIFT με παράνομο τρόπο, αλλά θα ήθελα να ξέρω αν αυτό έχει γίνει πριν ή μετά τον Ιούλιο του 2010. Εγώ χαιρετίζω ιδιαίτερα τη δική σας διαπίστωση που λέτε ότι μέχρι στιγμής έχουμε κάποιες καταγγελίες και κατηγορίες, δεν έχουμε όμως ε, αποδείξεις. Έχουμε διαψεύσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά καταρχήν είναι απαραίτητο να έχουμε όλα τα στοιχεία πάνω στο τραπέζι και να μπορέσουμε μόνο έτσι να καταλήξουμε σε μια πραγματική εκτέμηση. Δεν μπορούμε λοιπόν τώρα να καταλήξουμε στα συμπεράσματα όταν δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, να έχουμε πρώτα όλα τα στοιχεία μπροστά μας και μετά αφού κάνουμε την ε, εξέτασή τους να δούμε εάν χωρεί η προβληματική της καταγγελίας συμφωνίας ή όχι. Ευχαριστώ. Λάτφορντ. Προσεκτικά στο χρόνο. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ. Έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, έχω μάλλον για τις παρατηρήσεις σας. Θα ήθελα απλώς κάποια πράγματα. Η απάντηση του κυρίου Κοέν από το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρησιμοποιεί το TFTP για να έχει στοιχεία SWIFT που δεν μπορεί να έχει από άλλες πηγές. Δηλαδή δεν, αφορούν, δεν θεωρούν το TFTP ως ένα αποκλειστικό πλαίσιο για να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του SWIFT. Απλώς θεωρούν ότι είναι ένας βοηθητικός, μια βοηθητική δίωδος. Κατά τη γνώμη σας αυτό είναι παράβαση της συμφωνίας TFTP. Θεωρείτε ότι η συμφωνία TFTP είναι η μόνη νομική βάση για πρόσβαση στα στοιχεία του SWIFT. Είπατε εσείς ότι οι ισχυρισμοί αυτοί, αν είναι αλήθεια, θα ήταν, σημάνουν παραβίαση της συμφωνίας διότι υπό το άρθρο 1 της συμφωνίας τα στοιχεία που δίνονται προς το Υπουργείο Οικονομικών και μετά, όπως το καταλαβαίνω, που έπειτα μεταβιβάζονται στις αρχές επιβολής του νόμου ή αναχές τρομοκρατίας. Αλλά αυτά τα στοιχεία πάνε στην NSA είναι σωστά, είναι ακριβή. Τι σημαίνει δηλαδή αρχές ε, αντιτρομοκρατίας, ε, ε, επιβολή του νόμου, είναι και οι υπηρεσίες αντικατασκοπίας. Πάντα έχω αμφιβολία για την νομοθεσία. Αυτό είναι ένα κενό. Αν η NSA παίρνει τα στοιχεία από το δικό της Υπουργείου Οικονομικών, εντάξει. Αν τα παίρνει μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας TFTP, δεν εντάξει. Αυτό είναι το, το θέμα. Αυτό είναι... Άμα το παίρνει από το Υπουργείο Οικονομικών της, είναι σύμφωνο με την συμφωνία μας ή όχι. Προσπαθώ να καταλάβω. Ευχαριστώ κυρία Ρομέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Μάλμστρομ, επειδή είπατε στην παρέμβασή σας ότι εξηγήσει σας έδωσαν δεν σας ικανοποιούν, εξήγησε του κυρίου Κόεν. Τι ακριβώς αναμένετε να λάβετε ως εξήγηση από τις ΗΠΑ. Θα ήθελα να μου πείτε ακριβώς τι περιμένετε να σας εξηγήσουν για να θεωρείτε, θεωρήσετε ότι πλέον ε, είστε ικανοποιημένοι με την εξαγωγή αυτή τη συμφωνία που ήταν και ένα επίμαχο θέμα από την αρχή. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι ΗΠΑ μπορούν όχι μόνο με του Ευρωπαίου πολίτε ε, να κάνουν αυτά που κάνουν, αλλά και με του πολίτε όλου του κόσμου. Το θέμα είναι, έχει η Ευρώπη και σε ποιο βαθμό έχει μηχανισμού για να φρενάρει την ε, παρέμβαση αυτή στην ιδιωτική ζωή των πολιτών. Έχετε σκεφτεί ενδεχομένως να έχετε ένα είδος συνομιλίας ε, διαλόγου με την επιχείρηση SWIFT η επιχείρηση SWIFT υποχρεούται να δίνει στοιχεία στις κυβερνήσεις και των ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό που γίνεται με τις ΗΠΑ είναι ότι υποχρεούται να τους δώσει τα στοιχεία η επιχείρηση SWIFT. Αυτή η εταιρεία λοιπόν, αυτή η επιχείρηση υποχρεούται να δώσει στοιχεία και στις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό θα ήταν επίσης σημαντικό να το γνωρίζουμε για να δούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Γιατί αυτή τη στιγμή η κατάσταση όχι μόνο για τους Ευρωπαίους υπηκός αλλά και για τους υπηκός όλου του κόσμο είναι ότι ε, δεν είμαστε προστατευμένοι, είμαστε εντελώς απροστάτευτοι και δεν έχουμε καμία προστασία. Αυτά τα δημιουργεί ο νέος κόσμος στον οποίο ζούμε και διερωτώ με, τι μηχανισμούς έχει η Ευρώπη για να το αντιμετωπίσει αυτό. Διότι να είναι ο επόπτης η Ευρωπόλ δεν είναι κάτι το οποίο μας έψε και ποτέ γιατί πολλές φορές ήρθε και θα ξανάρθει αλλά εξηγήσει δεν θα λάβουμε και ο Ευρωπαίος Επόπτης Δεδομένων είπε και ο κύριος ε, ε, ότι θα πρέπει να βρούμε έναν ανεξάρτητο ETPS, έναν ανεξάρτητο επόπτη Όμω ε, όμως εμείς δεν έχουμε καμία τέτοια προσωπικότητα, δεν έχουμε καμία προσωπικότητα σε κανένα μηχανισμό και ακόμα πιο σοβαρό είναι ότι για τη διεθνή καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχουμε οδηγίες για αυτό. Δεν γίνεται λόγος για αυτό το θέμα καθόλου. Μόνο για τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ γίνεται λόγος. Και είναι πάρα πολύ πιο σοβαρό θέμα η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας παρά η απλή συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ, αλλά παρακαλώ να έχετε υπόψη σας ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Διάθετε μέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόνο σε μία ιδέα θα σταθώ. Να πω προηγουμένως όμως ότι εγώ κατανοώ απόλυτα αυτά τα οποία είπε ο Άξελ Βος και ο, και ενώ Σπίρκελ. Ενώπιόν μας τώρα έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και αμφιλεγόμενη. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την έννοια της ασφάλειας θα πρέπει να υπενθυμίσω το εξής. Η απόφαση του, η συμφωνία του Ιανουαρίου έχει και ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή. Συμφωνώ με την κυρία Μάλσομ σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία. Μου φαίνεται όμως κυρία Μάλσομ ότι έχει και ρήτρε στη συμφωνία που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν τέσσερις αμερικανικοί νόμοι που επιτρέπουν την προσφυγή στη δικαιοσύνη σε περίπτωση μη τήρησης της ε, συμφωνίας. Ο νόμος του Γενικού Επιθεωτή του 1978, ο νόμος της διοικητικής διαδικασίας του 1946 και τέλος ο νόμος για τις καταχρήσεις και τις απάτες στο διαδικτύο. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να προσφύγουμε στα αμερικανικά δικαστήρια. Επί τη βάση αυτών που αναφέρονται λοιπόν στη διαδικασία μπορούμε να ξεκινήσουμε μια διαδικασία στα αμερικανικά δικαστήρια. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και πάλι να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά ερωτήματα σε σχέση με το SWIFT και φυσικά αυτά τα προβλήματα και τα ερωτήματα υπήρχαν πολύ πριν ανακαλυφθούν αυτά τα οποία καταγγέλνουν οι πρόσφατες δημοσιεύσεις για το SWIFT. Η πρόσβαση λοιπόν της NSA στα δεδομένα του SWIFT. Αναφέρατε ότι υπάρχει ένα έγγραφο που δείχνει ότι μπορεί να το κάνει αυτό και νομίζω ότι είναι σαφές ότι μια μυστική υπηρεσία μπορεί να κάνει κάτι, θα το κάνει αργά ή γρήγορα. Επομένως, ποιος είναι αυτός ο οποίος ελέγχει κατά πόσο υπάρχει πρόσβαση ή όχι σε αυτά τα δεδομένα από την ευρωπαϊκή πλευρά και ποιος ελέγχει ότι χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς από την πάταξη της τρομοκρατίας. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι δεν είναι μονάχα οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι και άλλες πολλές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν σε μια φαιά περιοχή, στην οποία δεν υπόκεινται σε καμία απόλυτη, <clears throat> απόλυτα ε, εποπτεία και κανείς δεν μπορεί να διακριβώσει τι ακριβώς κάνουν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα με το να παγώσουμε αυτή τη συμφωνία. Αυτό είναι γελίο για μένα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία, όχι να την καταγγείλουμε. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία και να πείσουμε τον εαυτό μας ότι δεν γίνεται μια παραβίαση αυτής της συμφωνίας ή το αντίθετο. Και επίσης σε αυτά που είπε ο κύριος ε, Άλβαρο για την TFTP. Εγώ δεν είμαι απόλυτα σίγουρα, σίγουρη αν εμείς έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα δικό μας πρόγραμμα προστασίας των δεδομένων αν καταγγείλουμε αυτή τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ο κύριος Μέλντορ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω πως η προσέγγιση της Κομισιόν ήταν σωστή έχει θέσει τις σωστές ερωτήσεις, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι και ότι δεν θα λάβουμε ικανοποιητικές ε, ε, απαντήσεις. Και έπειτα θα πρέπει να επανέλθω σε αυτά που ήδη ανέφεραν συνάδελφοι, ότι αυτή τη στιγμή δίνουμε στοιχεία στις ΕΠΑ και πάνω κάτω τα κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε παρκώς, κατά τη γνώμη μου, και η μόνη λύση είναι να φτιάξουμε εμείς ένα είδος κέντρο που συλλέγουμε στοιχεία και που μόνο έπειτα από συγκεκριμένα αίτημα την είπα θα τα δίνουμε και όχι άντε μπάτε σκύλια λέστε να ρωτήσω λοιπόν από την Κομισιόν ποιες είναι οι προπτικές και οι δημοσιονομικέ να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο στην Ευρώπη και σύντομα υπάρχει κάποια σχετική προετοιμασία Υπάρχει δηλαδή τρόπο να συλλέγουμε εμεί εδώ τα στοιχεία και άμα έχουν κάποιο συγκεκριμένο αίτημα ή είπα, να μπορούμε να του τα δίνουμε ή μη, να αποφασίζουμε ένα περίπτωση. Ευχαριστώ κύριο Μπορκέτσιο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω το πλεονέκτημα να πάρω τελευταίο το λόγο, όπω πάντα. Όχι, δεν είστε ο τελευταίο. Όχι, έχει και άλλου δύο. Εντάξει, πάση περιπτώσει. Σχεδόν τελευταίο. Και πολλά ερωτήματα ήδη έχουν τεθεί. Το δικό μου ερώτημα είναι πολύ σύντομο και ξεκάθαρο. Κυρία, την οποία σέβομαι απόλυτα, αλλά εσείς ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν νομίζετε ότι έχετε κάνει μια ομιλία σαν να ήσασταν ηλίκοι στη χώρα των θαυμάτων. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνεται σαν... Ε, είναι μια ένωση ηλικιωμένων που πάνε για προσευχές το βράδυ. Ε, όλοι μαζί. Με το έσελον υποτίθεται ότι έχουμε προστασία για τα στοιχεία μας. Εσείς ποια εγγύηση χρησιμοποιήσατε συγκεκριμένα για να αποφύγετε όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν τον ιδιωτικό χώρο των Ευρωπαίων πολιτών, την οικονομία, τις επιχειρήσεις κτλ. Όλα αυτά να μην τεθούν σε διάθεση όσων μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ενάντια στα συμφέροντα των Ευρωπαίων. Εσείς αυτοί οι ελεγκτές, μιλήσετε για δύο ελεγκτές να μας δώσουν μια έκθεση για τα όσα έκαναν και έπειτα ή είναι ανίκατοι, ανίκανοι και πρέπει να απολυθούν είτε δεν έχουν τα νομικά και τεχνικά μέσα στη διάθεσή τους και άρα η ευθύνη είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η διαφάνεια που είναι, είναι αυτό το οποίο απαιτείται αυτή τη στιγμή θα πρέπει να φέρουμε άπλετο φως σε όλη αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το τεραστίων διαστάσεων σκάνδαλο. Έχουμε ακούσει όλες αυτές τις κατηγορίες, όλες αυτές τις ε, καταγγελίες. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να υπάρξει απόλυτη σαφήνεια για όλα αυτά. Επιπλέον, θέλω να πω το εξή. Από ό,τι φαίνεται, η NSA έχει τη δυνατότητα να συλλέξει στοιχεία προσωπικά Ευρωπαίων και κατά πάσα πιθανότητα το έχει πράξει, έχει λάβει, έχει πάρει στοιχεία ατόμων, επιχειρήσεων, τραπεζών και όλα αυτά έχουν γίνει με την κάλυψη της συμφωνίας που, έχει, που ισχύει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την συμφωνία αυτή έχει καταφέρει να έχει την ε, κτίση των στοιχείων αυτών. Αλλά υπάρχει και μία δεύτερη δυνατότητα που αναφέρεται στα μέσα ενημέρωσης ότι γίνονται πραγματικά παράνομες παρακολουθήσεις ή παράνομη απόκτηση στοιχείων πέραν και επέκεινα της συμφωνίας αυτής. Θα ήθελα να φέρω στο εξή ερώτημα. Μπορεί η Κομισιόν να εξηγήσει με σαφήνεια στους Ευρωπαίους πολίτες τι ακριβώς έχει συμβεί ή όχι. Θα πρέπει να φερω το ο Ευρωπαίος πολίτης να ξέρει τι γίνεται με τα δεδομένα του. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να ξέρουν, να ξέρουν οι πολίτες αυτοί προς ποιους σκοπούς θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά οι Ηνωμένε Πολιτείε. Εγώ πιστεύω ότι έχει υπάρξει μια παραβίαση, μια παράνομη διαδικασία και επομένως θα πρέπει να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την παραβίαση. Και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να πει κανείς απλώς ότι αφορά μονάχα ένα μικρό τμήμα Ευρωπαίων πολιτών ή ελάχιστες τραπεζικές ε, ε υποθέσεις, ελάχιστους τραπεζικούς λογαριασμούς. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν και μια, μια δικαστική διαδικασία γιατί πρόκειται για παραβίαση συγκεκριμένων ατόμων που έχουν παραβιαστεί. We can turn back to our Commissioner Malmström. Yes, right. Thank you. Um, do you suspect... Μάλιστα, ευχαριστώ. Υποψιάζεστε ότι η κατηγορία των στοχευμένων ε, ατόμων για τα, οποία, τα στοιχεία των οποίων ενδιαφέρεται η NSA ε, είναι μεγαλύτερος ο κατάλογος αυτός από αυτούς που είναι ύποπτοι για τρομοκράτες ή ε, για συμμετέχοντες σε οργανωμένο έγκλημα. Εξάλλου η ΙΠΑ δεν θεωρούσαν τρομοκράτες τον IRA ούτε και τους κόντρας στην Κεντρική Αμερική, ούτε και τους Ισλαμιστές ανάμεσα στην ε, Συριακή αντιπολίτευση. Άρα λοιπόν, ε, σε μια πρόσφατη ε, ακρόαση εδώ, ο κ. Applebaum, που ανησυχούσε ευρύτερα για την εποπτεία NSA, ισχυρίστηκε ότι οι ερευνητές δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί ακτιβιστές ε, επίσης κατηγοριοποιούνται ως τρομοκράτες. Πόσο ευρύ είναι το φάσμα των πολιτών που μπορούν, μπορεί νόμιμα και θεμητά να ερευνάται. Πού είναι το όριο των τρομοκρατών. Και στη φάση που διαπραγματευόμασταν την συμφωνία SWIFT, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θεώρησε ότι ότι οι όροι περί ασφαλείας θα ήταν πολύ σημαντική όρια για αυτή τη συμφωνία. Εφόσον αυτοί οι όροι έχουν παραβιαστεί, τότε ολόκληρη η συμφωνία έχει παραβιαστεί και άρα δεν έχουμε καμία υποχρέωση. Πρέπει απλώ να ανασταλεί, να ακυρωθεί. Και έπειτα, πώ ήταν δυνατόν οι ΗΠΑ να ξεπεράσουν τι ασφαλιστικέ δικλείδε ε, για την πρόσβαση σε στοιχεία. Αν αυτέ οι ασφαλιστικέ δικλείδε δεν μπορούν να εμποδίσουν τι ΙΠΑ από το να έχουν πρόσβαση, τότε έχουμε πρόβλημα με την ασφάλεια ή με τα άτομα που εφαρμόζουν την ασφάλεια. Ευχαριστούμε. Εσεί τώρα, κυρία Μάλστρομ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να μιλήσω, να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Άλμπρεχτ γιατί δεν απάντησα την ερώτησή του, γιατί είναι κάπως εκτός του πεδίου αυτό. Υπάρχουν δύο ομάδε εργασία, ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στο Συμβουλίο, που η Κομισιόν δεν έχει ρόλο να συζητήσει με διαφορετικές εικασίες ότι οι ΙΠΑ ε, ε, κρυφακούν στι πρεσβείε τις ευρωπαϊκές και έπειτα υπάρχει άλλη ομάδα εργασίας όπου ε, συμμετέχουν η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. Και εκεί σταδιακά προσπαθούμε να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα και κάποια έκθεση. Είναι κάπως νωρίς να πούμε τι θα προκύψει και επίσης ε, ε, περιμένουμε να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια. γι' αυτό θέλω να μιλήσω μόνο για το shift σήμερα και ξέρω ότι ο κ. το απόγευμα θα μιλήσει για το τα υπόλοιπα. Η Κομισιόν δεν σκοπεύει να φτιάξει ένα κέντρο δικατασκοπίας. Αυτό που θέλουμε, έχει προταθεί είναι η ένα είδος ευρωπαϊκού TFTP. Αυτό βεβαίως μπορεί να συζητηθεί για το κατά πόσο μπορούμε να το κάνουμε ή όχι, αν να το κάνουμε ή όχι και αυτό το εξετάζουμε στην ανακοίνωση που ετοιμάζουμε ότι δηλαδή αυτό έχει πολλές επιπτώσεις εάν θα είναι μόνο στοιχεία του SWIFT γιατί σήμερα τα χρήματα μεταφέρονται με πολλούς άλλους τρόπους υπάρχουν πολλοί τρόποι να μεταφέρει κανείς χρήματα να κάνει έμβασμα και αυτό θα πρέπει να συζητηθούν βεβαίως σε ευρύτερο πλαίσιο και όσον αφορά τι διάφορες αξιολογήσεις, αναθεωρήσεις ε, και τα λοιπά και την εποπτεία που έχουμε τους ελεγκτές. Μέχρι σε εμφανιστούν τα πρώτα άρθρα δεν είχαμε καμία απολύτως ένδειξη ότι υπήρχε παράβαση της συμφωνίας, παραβίαση μάλλον της συμφωνίας. Και βεβαίως όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί τους οποίους και εγώ διάβασα στα ΜΜΕ θα πρέπει να διευκρινιστούν και γι' αυτό και υπάρχουν ερωτηματικά πολλά αυτό το ερώτημα που έθεσε ο κ. Μπρόνς για το πεδίο εφαρμογής αυτό ορίζοντα το άρθρο 2. Τι εστί τρομοκρατία. Και φυσικά και αυτή η ερώτηση θα πρέπει να τεθεί. Αν το ξεπέρασαν αυτό, αν ήταν καθαρά για ε, αντιτρομοκρατικούς σκοπούς ή για σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων κτλ. Και γι' αυτό και υπάρχει και το άρθρο 2 στη συμφωνία όπου περιλαμβάνονται οι ορισμοί. Το, το ερώτημα της κυρίας Λάτφορντ είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, διότι εάν στοιχεία που βγαίνουν από, τα SWIFT, από το SWIFT σχετίζονται με μια συνεχιζόμενη έρευνα για την τρομοκρατία ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αφού τα έχουν εξετάσει τα δώσουν σε άλλη αρχή, αυτό είναι σύμφωνο προς τη συμφωνία εν Πρέπει κανείς να δει τις λεπτομέρειες. Αλλά αν η NSA άμεσα πήγε και πήρε ε, στοιχεία, τότε είναι κάτι τελείως διαφορετικό και συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει αυτό να διευκρινιστεί. Τι ακριβώς έγινε δηλαδή. Το ένα σημαίνει παραβίαση, το άλλο όχι. Είναι το πρώτο και κύριο ερώτημα που πρέπει να τεθεί. Αυτό πρέπει λοιπόν ε, ίσως να το διευκρινίσουν οι συνάδελφοι από τη ΣΥΟΥΦΤΗ και το Γεροπόλε για να, τα πιο τεχνικά θέματα, τα πολιτικά ζητήματα που σχετίζονται με τους ισχυρισμούς, ε, τις καταγγελίες και τη συμφωνία. Νομίζω τα απάντησα, θα σταθώ σε αυτά και φυσικά επαναλαμβάνω την διαθεσιμότητά μου. Εγώ και οι υπηρεσίες μου ε, να ερχόμαστε τακτικά να συζητάμε αυτά τα θέματα. Πράγματι, όπως σας είπα θα έχουμε και τον κύριο Wainwright από την Europol και την κυρία Πλάνς Πέτχα στην επόμενη συνεδρία μας. Είναι εκπρόσωπο ε, του Συμβουλίου τη εταιρεία SWIFT, τη εταιρεία την οποία συζητάμε, αλλά πρώτα απ' όλα να μα πει λίγα πράγματα ο κ. Ντεμπόκελε από την ε, Βελγική Αρχή Προστασία Δεδομένων, τη Belgacom. Δεν ξέρω αν είναι εδώ ο κ. Ντεμπόκελερ, είναι εδώ. Μάλιστα. Σας καλέσαμε. Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια, αλλά θα ήθελα να εστιάσετε δυνατόν στην υπόθεση SWIFT. Και όπως αναφέρθηκε στα διάφορα δημοσιεύματα οι ε, πληροφορίες που οδήγησαν και στην όλη αυτή εξεταστική διαδικασία, τι γίνεται με την υπόθεση SWIFT συγκεκριμένα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο ε, σε ό,τι αφορά το SWIFT. Όταν μετά τις 25 Ιουνίου 2006 φάνηκε ότι το SWIFT ε, ερευνά το ε, γενικώ από τις ε, υπηρεσίε ε, πληροφοριών ασφαλείας των ΙΠΑ αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών ε, οι οποίοι ουσιαστικά ερευνούσαν όλες τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και μετά από μήνες συζητήσεων στις 8 Δεκεμβρίου του 2008 βρέθηκε μια συμφωνία, ένα settlement μεταξύ της αρχής, της Προστασία Αρχής Προστασίας Δεδομένων και της εταιρείας SWIFT. Με βάση αυτή την συμφωνία, η εταιρεία SWIFT ενέκρινε μέτρα τα οποία θα επέτρεπαν την προστασία της πελατείας της και των χρηστών του δικτύου της. Εξασφαλιζόταν δηλαδή γενικά η προστασία των πολιτών. Υπήρξαν τρεις ε, συναντήσεις ε, παρακολούθησης ε, από το 2008 και μετά. Εμείς, η Βελγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, ελέγξαμε την εκτέλεση των μέτρων, την εφαρμογή των μέτρων αυτών και μέχρι στιγμής συστηματικά διαπιστώνουμε ότι οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η εταιρεία ΣΥΕΦ το 2008 τηρούνται στην πράξη. Και σε αυτό το πλαίσιο δεν διαπιστώσαμε και κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στον τομέα της επεξεργασίας ε, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών. Υπάρχει όμως ένα δεύτερο κύκλωμα παρακολούθηση, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, στο πλαίσιο της συμφωνίας τη FTP και έχουμε μια κοινή ομάδα αξιολόγηση μεταξύ ΙΠΑ ΕΕ, το αναφέραμε αυτό, και είναι και αντικείμενο δύο εκθέσεων ήδη. Ούτε όμως αυτό το πλαίσιο εντοπίσαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων. Η Επιτροπός Μάλστρομ ήδη το είπε. Εξετάζονται επίσης ε, και οι εργασίε της Europol από την κοινή αυτή ομάδα, νυχτή ομάδα αξιολόγηση. Εντοπίστηκαν κάποια προβλήματα εδώ όμως, ιδίως στον ε, τομέα της κατανόησης και της εφαρμογής ε, της συμφωνίας τη FTP. Και ιδίως όταν ε, η μεταφορά δεδομένων γίνεται χίδινη όχι αν θέλετε. Σε ό,τι αφορά το SWIFT, το μόνο που μπορώ να σας πω τελικά είναι ότι στο παρόν στάδιο δεν έχουμε ενδείξεις ή αποδείξεις που να μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε ε, την ύπαρξη προβλημάτων σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Ντεμπερκλερ. Ξέρουμε ότι σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες για παράνομη πρόσβαση στα συστήματα της Belgacom ότι και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συνδέεται με την υπόθεση της SWIFT και πιστεύω ότι θα έχουμε και περαιτέρω ευκαιρίες να συζητήσουμε το θέμα αυτό γιατί τις 3 Οκτωβρίου θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, όπως έχει ανακοινωθεί. Και να μην καθυστερήσουμε περισσότερο, λοιπόν, θα ήθελα να δώσω το λόγο στο, Wayne, στο Rob Wainwright, τον διευθυντή της Europol, για να μας παρουσιάσει τις απόψεις του για το θέμα αυτό. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε από την κυρία Μπλόνς Πέτρε για τα θέματα SWIFT και θα συνεχίσουν και πάλι ανταλλαγές ερωτήσεων αλλά και απαντήσεων. Κύριε Wainwright. Α, σας έψαχνα. Είστε απόλυτα καλό δεκτός για να λάβετε το λόγο και να μας παρουσιάσετε τις απόψει. σας. Ευχαριστώ. Εάν θέλετε να έρθετε εδώ πέρα. Είσαστε και οι δύο απόλυτα καλόδεκτοι να έρθετε στα προεδρικά θεωρία, ώστε να είσαστε και ορατότεροι morning. Of course. The floor is yours. Έχετε το λόγο. <clears throat> Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους και όλους. Χαίρομαι λοιπόν που έχω την ευκαιρία να κάνω ενώπιον σας κάποιες σύντομες παρατηρήσεις από τη Europol για το συγκεκριμένο αυτό θέμα και τις έρευνες που έχουν να κάνουν με τις καταγγελίες ότι η NSA έχει παράνομη πρόσβαση στα δεδομένα της ε, SWIFT. Δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα σε αυτά που είπε η κυρία Μάλστομ για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα αυτά. Είναι απόλυτα στην Κομισιόν φυσικά σε θεσμικό επίπεδο να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Η Ευρωπόλ δίνει ως το περισσότερη υποστήριξη, αλλά προς το παρόν, όπως είπε και η κυρία Μάτσομ, προσπαθούμε να εξετάσουμε το τεχνικό έργο της εφαρμογής αυτών των τμήματων της συμφωνίας, για τα οποία έχει αρμοδιότητα η Europol. Η Europol βέβαια είναι πάντα έτοιμη να υποστηρίξει αυτή την έρευνα με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι σημαντικό όμως να αναφέρω ότι υπάρχουν και κάποιοι εθνικοί περιορισμοί εγώ δεν μπορώ να εκπροσωπήσω την άποψη των υπηρεσιών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε ένα όργανο επιβολής του νόμου, δεν είμαστε <clears throat> υπηρεσία πληροφοριών. Μας απασχολεί το διεθνές ε, ε, υπερεθνικό έγκλημα και η τρομοκρατία. Βέβαια, συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για τις εθνικές διοκτικές και δικαστικές δυνάμεις και έχουμε μια περιορισμένη εμπειρία συνεργασίας με υπηρεσίες ασφαλείας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας επί τη βάση δήλωσης του 2004 μετά από την τρομοκρατική επίθεση στην ε, Μαδρίτη οδήγησε στη δημιουργία μιας ειδική μονάδος στην Europol με στόχο να ενθαρρύνει περισσότερο την συνεργασία μεταξύ της Ευρωπόλ και των υπηρεσιών ασφαλείας. Έχουμε λοιπόν την δυνατότητα αυτή. Όλα τα... Όλα αυτά τα δεδομένα υπόκειται στην γνωστή στην Επιτροπή σας διαδικασία προστασίας δεδομένων που είναι ιδιαίτερα στεναρή και ισχυρή. Αυτό ανεξάρτητα από την ε, προέλευση αυτών των δεδομένων. Η νομοθεσία αυτή ε, διέπει και τις σχέσεις Europol με τις εθνικές αρχές και βέβαια η Ευρωπόλ δεν μπορεί να συλλέξει ή να αποθηκεύσει δεδομένα τα οποία έχουν αποκτηθεί με παράνομο τρόπο ή που δεν συνάδουν με την νομοθεσία των χωρών μελών. Όλες οι πληροφορίες λοιπόν αυτού του είδους ε, δίδονται επί τη βάση της εθνικής νομοθεσίας στα κράτη-μέλη για όλες τις χώρες με τις οποίες έχουμε μια συμφωνία. Είναι βεβαίω ακόμα δυνατόν μέσα στο πλαίσιο νομικό που ισχύει κάποια στοιχεία που λάβαμε με αυτόν τον τρόπο η Europol να προκύπτουν από τα αντίστοιχε υπηρεσίες τι αστυνομικέ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του εκάστοτε κράτους μέλου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ε, έχουν ε, δοθεί στην Europol με συγκεκριμένο τρόπο ε, έτσι ώστε η Europol να μην μπορεί να εντοπίσει την ε, πραγματική πηγή αυτού του υλικού. Βέβαια θεωρώ πως μόνο ένα μικρό ποσοστό των στοιχείων αυτών που προκύπτει από τις υπηρεσίες αντικατασκοπίες είναι ε, κατά παραγγελία. Τα υπόλοιπα προκύπτουν από τις εργασίες των αστυνομικών αρχών. Τώρα, ε, ρυθμίσεις συνεργασίας έχουν θεσπιστεί με διάφορες ε, υπηρεσίες επιβολής του νόμου των ΙΠΑ. Ορισμένες έχουν μάλιστα εκπροσώπους στα δικά μας αρχηγεία, για παράδειγμα. Και το τελευταίο μήνα αυτή η συνεργασία οδήγησε σε 50 επιχειρήσει διεθνούς ε, ε, φύση. και εδώ καλύπτεται το πλήρε φάσμα σοβαρών διεθνών εγκλημάτων. Στον τομέα των ε, στοιχείων αυτών και πάλι έχουμε στοιχεία μόνο από τις ε, υπηρεσίες ε, επιβολής του νόμου. Δεν έχουμε καμιά επαφή με την NSA ούτε με τη CIA. Ανταλλαγή πληροφοριών με τη ΣΥΠΑ ε, φυσικά καλύπτεται από τις ίδιες εντολές και εγγύησεις που καλύπτει και η, καλύπτεται και η εργασία της Europol. Ε, λογικότητα ας πούμε εφαρμόζεται όπως και στην περίπτωση εργασίας, συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Επίσης είναι πιθανόν στη θεωρία κάποιες από τις πληροφορίες της Europol να προκύπτουν από τις ε, από την NSA ή από άλλες ε, ε, αρχές των ΙΠΑ, αλλά δεν είναι και τόσο πιθανό λόγω της περιοριστικής ερμηνείας ε, της συνεργασίας, της συμφωνίας μάλλον συνεργασίας μεταξύ Europol και ΙΠΑ, που οι ΙΠΑ εφαρμόζουν και εμποδίζουν τις διαβαθμισμένες πληροφορίες. Μάλλον ε, ε, βάζουν φραγμούς για την μετάδοση των ε, διαβαθμισμένων πληροφοριών. Έτσι ερμηνεύει την νομική τη συμφωνία η Αμερικανική Αρχή. Δεν μοιράζεται πληροφορίες με το Europol εκτός από το συγκεκριμένο πλαίσιο της συμφωνίας TFTP. Αυτό σημαίνει ότι οι δικές μας γνώσεις της NSA και της αντικατασκοπίας των ΙΠΑ ε, είναι πολύ χαμηλή, πολύ αμυδρή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ευρύτερη συζήτηση, σε σχέση με τις δραστηριότητε της NSA, εμείς δεν συνεργαζόμαστε με την υπηρεσία αυτή και δεν έχουμε κάποιο ιστορικό του να παίρνουμε πληροφορίες από την NSA ή τουλάχιστον που γνωρίζουμε ότι προέρχονται από εκεί σε σχέση με την ίδια τη συμφωνία TFTP. Δεν έχω να σας πω τίποτα περαιτέρω αυτό που σας είπε η Επίτροπος Μάλστρομ. Φυσικά είμαι υπεύθυνος για να εξασφαλίσω ότι είναι και αυτή απόλυτα πληροφορημένη από την Europol. Αν είχαμε κάποια στοιχεία τα οποία ερχόντουσαν σε αντίθεση με αυτά που, θα σας, που σας είπε η κυρία Μάλστρομ, θα την ενημέρωνα. Η οργάνωση των ανταλλαγών δεδομένων Ε, γίνεται με τον ίδιο τρόπο που σας παρουσίασε η κυρία Επίτροπος. Εμείς βέβαια θα παραμείνουμε πιστοί στον ε, επιχειρησιακό μας στόχο όπως με επακριβή τρόπο περιγράφεται στη συμφωνία TFTP. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση TFTP έχουμε φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο για την ε, εφαρμογή των διατάξεων αυτών από εμά, παρά το γεγονό ότι είναι πολύπλοκο το έργο αυτό και επίσης ε, φαντάζομαι ότι το θέμα της σημασίας και της αξίας αυτής της συμφωνίας δεν είναι απόκειται σε μένα να το κρίνω. Είναι καλό να σας πενθυμίσω όμως ότι αυτή η συμφωνία ε, καλύπτεται και από την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου ε, προστασίας δεδομένων και τον πλήρη έλεγχο από το κοινό εποπτικό μας φορέα και όλες τις άλλες διασφαλίσεις. Η Europol έχει πάντα συνεργαστεί με του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, αλλά δεν έχουμε καμία επαφή με μέλη της CIA ούτε της NSA ή τουλάχιστον με άτομα τα οποία γνωρίζουμε ότι ανήκουν σε αυτούς τους δύο ευαγείς φορείς. Και για να επαναλάβω αυτά που είπε η Κομισιόν, σε λειτουργικό επίπεδο αυτοί οι αξιωματούχοι πάντα υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία που παίρνουν οι Αμερικανοί από τη συμφωνία TFTP δεν προέρχονται από άλλες πηγές, έχουν σαν αποκλειστική πηγή λοιπόν οι πληροφορίες τους στην TFTP. Δεν έχουμε λοιπόν πληροφορίες που να δείχνουν ότι η NSA έχει, πρόσφατη, <clears throat> έχει μάλλον άμεση πρόσβαση στην SWIFT λόγω του τρόπου με τον οποίο, με τον οποίο λειτουργούμε θα ήταν απίθανο να ξέρει κάτι τέτοιο η Europol, αλλά σας λέω ότι δεν έχουμε πληροφορίες οι οποίες είτε να επιβεβαιώνουν είτε να διαψεύδουν τις πληροφορίες σε σχέση με την αποκτήση στοιχείων από την NSA. Επομένως, εν κατακλείδη. Η συμφωνία TFTP έχει σαν στόχο τον αγώνα κατά του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Διοκτική Αρχή δεν έχουμε άμεση επαφή με την CIA και την NSA. Έχουμε κάποια εμπειρία με τη συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών με τα κράτη-μέλη και μόνο αυτό είναι. Όλες οι ανταλλαγές δεδομένων της Europol υπόκειται στο πλαίσιο για τη διαβίβαση δεδομένων. Ενδεχομένως κάποια από τα στοιχεία τα οποία Εμεί ε, περνάνε από τα χέρια μας, προέρχονται από τι υπηρεσίε πληροφοριών, αλλά πάντα προστατεύεται η πηγή του όταν περνάνε τα κανάλια τη Europol και νομίζουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό των δεδομένων που έχουμε στα χέρια μα. Η Επιτροπή σας βέβαια κάνει μια έρευνα που την υποστηρίζουμε απόλυτα, όσο και το σημαντικό έργο της Κομισιόν να ζητήσει περισσότερα στοιχεία από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών και είμαι στη διάθεσή σας να βοηθήσω την Επιτροπή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γουένραιτ. Θα έλεγα τώρα ότι είναι μια καλή να ακούσουμε την κυρία Πέτρα. Παρακαλώ. Και μετά θα έχουμε ρωτήσει και απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που δίνετε στη σου τη δυνατότητα να μιλήσουμε σήμερα μαζί σας εδώ στην Επιτροπή σας τις ευθύνε μα στον τομέα τη φυσική δεδομένων τις αναλαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά ε, και αναγνωρίζουμε και το έργο τη επιτροπή σα ότι αφορά την προστασία δεδομένων. Ω εταιρεία εστιάζουμε βέβαια στην ασφάλεια την προστασία των δεδομένων και επομένω συμφωνούμε πάρα πολύ και συμμεριζόμαστε τι ανησυχίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στηρίζουμε τη δουλειά του και με τα χαρά θα συνεργαστούμε όσο περισσότερο μπορούμε με το Κοινοβούλιο. Θα πρότεινα λοιπόν πρώτα απ' όλα να σας ε, δώσω έτσι μια σύντομη επισκόπηση της εταιρείας μας ε, SWIFT και μετά θα αναφερθώ στα ζητήματα της ασφαλείας, της ασφάλειας στο SWIFT και της ασφάλειας του συστήματος τη Συμφωνία TFTP. Πρώτα απ' όλα για το SWIFT, όσοι δεν γνωρίζετε, η SWIFT είναι μια μεσαίου μεγέθους ε, ιδιωτική εταιρεία με την έδρα της εδώ στο Βέλγιο η οποία συστάθηκε το 1973 ως συνεταιρισμός. Στόχος ε, της SWIFT ήταν να αντικαταστήσει την Telex ε, και να ε, διευκολύνει την ασφαλή ανταλλαγή χρηματοοικονομικών μηνυμάτων μεταξύ χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Μετά λοιπόν από όλα αυτά τα χρόνια, τα 48 χρόνια λειτουργίας μας, η ασφάλεια και η προστασία είναι στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας μαζί με την εμπιστευτικότητα ε, των στοιχείων των πελατών μας. Και αυτές είναι οι προτεραιότητες μας υπηρεσίες παρέχουμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα και πάλι παραλαμβάνω ότι είμαστε ένας ε, πάροχος δεδομένων, δεν είμαστε τράπεζα, δεν είμαστε γραφείο συμψηφισμού για καθαρίσεων, παρέχουμε υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ εχματοπιστωτικών οργανισμών ε, και συνεταιρισμών. 10.000 είναι σήμερα οι πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυό μας. Πολύ σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε λογαριασμούς ε, και δεν δίνουμε πρόσβαση ή τέλο πάντων οι ιδιώτε δεν έχουν πρόσβαση και δεν μπορούν να επιλέξουν το σύστημά μα. Το σύστημά μα το χρησιμοποιούν μόνο χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί σε πάνω από 200 χώρες ε, ασκούμε την δραστηριότητά μα και δεν είμαστε όμω πάροχος υπηρεσιών, αλλά είμαστε και ένα φορέα τυποποίηση για την κοινότητα, για το χρηματοοικονομική ε, κοινότητα, το χρηματοοικονομικό κλάδο και αυτό το οποίο κάνουμε επίση είναι ότι παράγουμε κάποια υποδείγματα, templates ε, για το BIC ή για το SWIFT, τον κωδικό BIC, κωδικό SWIFT θα έχετε ακούσει φαντάζομαι και αυτά τα templates μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα πρότυπα όχι μόνο για το SWIFT αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο δίκτυο μέσω επικοινωνία. Αυτά για το SWIFT, πολύ γρήγορα έτσι περιεκτικά και συνοπτικά. Τώρα, ασφάλεια στο πλαίσιο του συστήματος SWIFT. Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ε, στο άλλο δυνατό επίπεδο προστασίας ε, και ασφάλειας ε, με βάση τα ισχυρά πρότυπα και επαναλαμβάνω ότι το, στο ότι κάνουμε κλειδί ε, είναι η προστασία των δεδομένων. Είναι ο πυρήνας της αποστολής μας ε, να έχουμε διαθεσιμότητα, εμπιστευτικότητα, ακαιρεότητα για τα δεδομένα των πελατών μας. Και έχουμε μηδενική ανοχή σε συμβάντα ε, που έχουν να κάνουν με τη διαθεσιμότητα ή την εμπιστευτικότητα ή ασφάλεια λοιπόν στο επικέντρο των δραστηριοτήτων μας. Άρα αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό για τους πελάτες μας. Αν εμπιστεύονται οι πελάτες μας ε, τη SWIFT, το κάνουν γιατί μπορούμε να τους παρέχουμε ασφαλείς υπηρεσίες. Και επενδύουμε και επανεπενδύουμε συνεχώς, διαρκώς, ε, για να είμαστε πάντοτε ε, έτοιμοι να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή μας το ανώτατο δυνατό επίπεδο και ιδίω γνωρίζοντα ότι κινούμαστε σε ένα πεδίο ε, απειλών. Δεν είμαστε λοιπόν ε, αυτάρισκοι σε καμία περίπτωση, δεν επαναπαυόμαστε. Να σα δώσω τώρα κάποια στοιχεία ό,τι αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά που έχουμε εφαρμόσει στο σύστημά μα. Έχουμε και λογικούς και φυσικούς ελέγχους. Πρώτος έλεγχος ασφάλειας είναι η κρυπτογράφηση είναι κρυπτογραφημένα τα μηνύματα SWIFT και έχουμε και πολλαπλά επίπεδα κρυπτογράφησης. Χρησιμοποιούμε την τελευταία τεχνολογία στον τομέα της κρυπτογράφησης. Κρυπτογραφούνται λοιπόν ε, τα μηνύματά μας από τη στιγμή που θα μπουν στο σύστημα μέχρι τη στιγμή που θα βγουν από αυτό, από το σύστημα SWIFT δηλαδή. Και όσο είναι αποθηκευμένα, τα μηνύματα είναι ε, κρυπτογραφημένα. Έχουμε επίσης ε, ένα πολλαπλό, ε, μια πολλαπλή δέσμη τείχων προστασίας, ε, firewalls, και είναι πολύ ε, προστατευμένα, θωρακισμένα θα έλεγα από τις απειλές της εσωτερικής και της τα μηνύματά μας ε, χάρη σε αυτά τα τείχη ασφαλείας. Επίσης δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το ε, δίκτυό μας δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είναι το περιβάλλον προστασία μας εντελώς απομονωμένο, stand alone, καμία πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και επίση έχουμε ενωπημένο σωματοποιημένου δασμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σύστημα εντοπισμού ανείχνευση για την ανείχνευση εισβολών. Έχουμε ένα τέτοιο σύστημα για να προστατεύσουμε την ακυριότητα του συστήματός μας. Έχουμε επίσης ε, κάποια ε, μηχανισμούς για να δούμε, να μελετήσουμε την ε, το ενδεχόμενο ε, εισβολών και ε, αξιολογούμε συνεχώς και προσωμιώνουμε τις απειλές. Έχουμε ένα πρόγραμμα επίσης ε, δοκιμής των παραβιάσεων, ή διεισδύσεων στο σύστημα, ώστε να μπορέσουμε σε περίπτωση που ανοιχνεύσουμε κάτι να αναλάβουμε αμέσως αποτελεσματική δράση. Έχουμε επίσης κατευθυντήριες γραμμές σε ό,τι αφορά τα δεδομένα τα οποία ε, πλέον δεν χρειάζεται να τα φυλάσσουμε για τη διάθεση αυτών των δεδομένων, για την απόρριψή τους, ώστε να μην μπορούν να ανακτηθούν αυτά τα δεδομένα. Υπάρχει επίσης ε, πάρα πολύ μεγάλος έλεγχος ό,τι αφορά το, το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνουμε και εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχουμε τα ε, χαρακτηριστικά του προσωπικού μας, το οποίο αποκτά έγκριση ασφαλείας και φυσικό έλεγχο, φυσικά υπάρχει και μέσα στο, στο επιχειρησιακό μας κέντρο πάρα πολύ αυστηρή είναι η πρόσβαση στους υπολογιστές μας. Ε, χρησιμοποιούμε ε, προσωπική αναγνώριση ταυτότητα, βιομετρικά στοιχεία, ε, χρησιμοποιούμε tokens και γενικά μπορούμε να ελέγξουμε πάρα πολλού τρόπου ε, αν κάποιο είναι εξουσιοδοτημένο ή όχι. Και φυσικά ελέγχουμε. Ελέγχουμε συνεχώ την ε, ροή δεδομένων στα συστήματά μα. Γνωρίζουμε ότι η κυβερνοαπειλές είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται, γίνεται όλο και πιο ε, συγκεκριμένο, επιτεδευμένο. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε, να ελέγχουμε τις ε, απειλές ε, και τα τροτά σημεία του συστήματος και να συνεχώς αξιολογούμε τους κινδύνους όπου τους, εντοπίζουμε και προσπαθούμε να εξελίσσουμε συνέχεια τα συστήματά μας και κάνουμε επίσης και κυβερνοασκήσεις για να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης. Είπα λοιπόν ότι η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της όλης μας αποστολής. Γι' αυτό και η ασφάλεια υπόκειται και σε εξωτερική αξιολόγηση. Η πρώτη σημαντική αξιολόγηση γίνεται από Τις κεντρικές τράπεζες οι οποίοι μας εποπτεύουν, ελέγχουν το SWIFT για να δουν ότι έχουμε πράγματι τις κατάλληλες διαδικασίες και τεχνικούς ελέγχους ε, ώστε η προστασία των δεδομένων να είναι μόνιμη. Η Εθνική Τράπεζα ε, του Βελγίου είναι βέβαια βασικός φορέας αφού είμαστε δηλωμένοι εδώ, αλλά και η ΕΚΤΑ είναι ένας από τους επόπτες μας, αλλά και η ΦΕΝΤΑ και η Τράπεζα της ε, Αγγλίας. Οι δέκα μεγάλες λοιπόν κεντρικές τράπεζες. Φυσικά έχουμε και εσωτερικούς ελέγχους, αλλά πέραν αυτού υποβαλόμαστε και σε ανεξάρτητους εξωτερικούς ελέγχους και τηρούμε τα διεθνή πρότυπα αναγνώρισης και σε αιτήσια βάση εκδίδουμε έκθεση με βάση τα ε, διάφορα πρότυπα. Συνοπτικά σας ανέφερα του έλεγχου ασφαλείας που έχουμε. Βέβαια δεν είναι πλήρης ο κατάλογος. Όπως σας είπα, συνεχώς ε, αναθεωρούμε και επανεξετάζουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας και προσθέτουμε νέους ελέγχους, νέα χαρακτηριστικά για να μπορούμε να εντοπίσουμε οποιαδήποτε μη εξωσιοδοτημένη χρήση. Όπως όλοι σας, έτσι και εμείς λοιπόν, διαβάσαμε τις πρόσφατες, ε, ε, τα πρόσφατα δημοσιεύματα, τους πρόσφατους ισχυρισμού. Και όλους αυτούς τους ισχυρισμού και τις καταγγείλεις αυτές τις λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Έχουμε τα μέτρα ελέγχου, τα μέτρα επαλήθευση. και σήμερα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχουμε ένδειξη ή απόδειξη ως προς το ότι υπήρξε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυό μας ή στα δεδομένα μας. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, πραγματικά θα μας είχε ανησυχήσει υπερβολικά. Και να είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε οποιαδήποτε κυβερνοαπειλή και αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει κίνδυνο στην ασφάλεια των υπηρεσιών μας, θα ερευνήσουμε πάρα αυτά και θα προβούμε πάρα αυτά στις ε, σκόπιμες δράσεις για να μετριαστεί αυτός ο κίνδυνος. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του SWIFT, της εταιρεία και του συστήματος SWIFT. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω εν συντομή για την ε, συμφωνία TFTP και γενικώ για τα αιτήματα ε, δεδομένων, χωρίξης δεδομένων. Ως η δυτική εταιρεία SWIFT φυσικά μπορεί να ε, λάβει αιτήματα, νόμιμα αιτήματα ε, για δεδομένα. Το 1993 είχαμε μια πολιτική συμμόρφωση σε ό,τι αφορά τα αιτήματα από τις αρχές των χωρών για δεδομένα. Το Συμβούλια όλων των ε, πελατών μας τα έχουν συζητήσει και εγκρίνει τα σχετικά αυτά και έχουμε και ένα λεγόμενο εγχειρίδιο χρηστών που περιλαμβάνει τις σχετικές διατάξεις και μπορεί να το βρει κανείς και στην ιστοσελίδα μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σας πω ότι πραγματικά ε, λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο ώστε να εξασφαλίσουμε το μίστο δυνατό προστασίας εμπιστευτικότητας, ακαιρεότητας, διαθεσιμότητας. Έχουμε νομικά δεσμευτικά αιτήματα από τις αρμόδιες αρχές τα οποία πρέπει να ανταποκριθούμε. Όταν λοιπόν και εφόσον μας ζητηθεί να παράσχουμε δεδομένα στις αρχές, αυτό το πράττουμε σεβόμενοι τις σχετικές συμφωνίες, αλλά και έχουμε μια πολιτική ώστε να εξασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων των πελατών μας. Ε, και γι' αυτό και οι αρχές γνωρίζουν τις βασικές αρχές προστασίας δεδομένων που διέπουν ε, ε, την εταιρεία. Αν λοιπόν ζητηθεί να δώσουμε στοιχεία, ε, προβαίνουμε, μάλλον εφαρμόζουμε την πολιτική μας ακριβώ και ο Επίτροπος νομίζω δεδομένων, προσωπικών δεδομένων του Βελγίου το 2008 αναγνώρισε αυτή την προσέγγισή μας. Τα μηνύματα SWIFT είτε έχουν μεταφερθεί ε, στο σύστημά μας, είτε όχι μπορούμε να, ε, μπορούν κάποιοι να τα λάβουν. Τώρα για το TFTP. Okay, thank you. So we, we... Είδατε ότι στη συμφωνία TFTP προβλέπονται ασφαλιστικές δικλείδες. Πέραν αυτών των ασφαλιστικών δικλείδων, εμείς ως επιτόπου εκπρόσωπος ε, και για να επαληθεύσουμε όλες τις ε, έρευνες ε, έχουμε τους δικούς μας ελεγκτές ανεξάρτητους, δεν θέλουμε να υπάρχουν παραθυράκια ή πισωπόρτες στο σύστημά μας και γι' αυτό μπορώ σήμερα να σας επιβεβαιώσω ότι δεν έχουμε κανένα απολύτως λόγο να πιστεύουμε ότι υπήρξε οποιαδήποτε μίξωση οδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα TFTP. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, δεν έχουμε καμία ένδειξη που να ε, δείχνει ότι ποτέ υπήρξε μη εξοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημά μας στα δεδομένα μας. Διατηρούμε την προστασία δεδομένων ε, ως προτεραιότητα, γιατί η εμπιστοσύνη στο σύστημα είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα συνεχίσουμε να συμμορφωνόμεθα προς, προς την νομοθεσία, αλλά επειδή η δραστηριότητά μας είναι παγκόσμια, και είναι ανταγωνιστικό το πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε σήμερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό η SWIFT να μην βρεθεί στη μέση. Γι' αυτό εκτιμώ τι προσπάθειε του Κοινοβουλίου, το οποίο σεβόμαστε και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας σε αυτό το πολύ σημαντικό ε, μέτωπο της προστασίας των δεδομένων. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πέτρα, λέει ο Πρόεδρος θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε πριν με την Επιτρόπο Μάλσον. Δηλαδή πρώτα θα μιλήσουν οι συγητές, μετά οι σκιώδεις και θα υπάρξει και ένας δεύτερος γύρος για τους υπόλοιπους βουλευτές που θέλουν τον λόγο. Επαναλαμβάνω και επιμένω δύο λεπτά ο καθένας. Διότι έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας και δεν έχουμε λίγους στον κατάλογο. Ξαναξεκινώ λοιπόν με τον εισηγητή κύριο Μωράης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω καταρχήν ότι οι σκιώδεις ρώτησαν για τους ισχυρισμούς του EASFGC που είναι το θέμα της συζήτησης για τις 3 Οκτωβρίου που έχουμε καλέσει εκπροσώπους από την ε, Βρετανία και από την Κόμμα. Ε, αυτό θα είναι το θέμα της συζήτησης ε, της 3 Οκτωβρίου όπως είπα. Τώρα για την εισήγηση του Rob Wainwright. Εάν κατάλαβα καλά, δεν ξέρω τώρα τι καταλάβανε οι υπόλοιποι, η Europol έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο υπό τη συμφωνία του 2010 και βασικά είπατε κύριε Γουένιράιτ ότι δεν γνωρίζατε καθόλου τι κάνουν η NSA και η CIA. Οπότε βασικά δεν γνωρίζετε ποιες είναι, ποιοι είναι οι ισχυρισμοί καταγγελίες. Εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να συνεχίσουμε να σας πιέζουμε. Τώρα δεν ξέρω πόσο θέλω πραγματικά να πιέσω έναν ανώτατο αστυνομικό, Βρετανό αστυνομικό. Αν θέλετε μπορώ και να το κάνω. Τώρα, εσείς μπορείτε να σχολιάσετε τι θα είναι μια αποτελεσμα... ποια θα ήταν μια αποτελεσματική δομή για την εποπτεία αυτής της συμφωνίας και έπειτα ποιο... πώς βλέπετε το ρόλο της Europol γιατί πολλοί κόσμος έχει περάσει χρόνο στη συμφωνία SWIFT για τη συμφωνία SWIFT και φυσικά σεβόμαστε την θέση της Europol εδώ αλλά έχετε ένα συγκεκριμένο ρόλο που αυτή τη στιγμή αμφισβητείται αυτό είπατε, ότι δεν γνωρίζετε καν ε, ποιες, είναι οι ισχυρισμοί. Ένα σχόλιο λοιπόν γι' αυτό και ένα σχόλιο για το μέλλον. Για το SWIFT, μπορώ να σας ρωτήσω και ξέρω ότι πρέπει να τα πείτε έτσι πολύ προσεκτικά. Πάντως η έκθεση στην Washington Post λέει ότι η ε, NSA από το 2006 παίρνει, σχολιάζει και χρησιμοποιεί τα στοιχεία Παρά λοιπόν ε, τις διάφορους κώδικες ε, κρυπτογραφήσεις ε, και τείχους, φραγμούς, τα χρησιμοποιούν μια χαρά. Τι μπορείτε να μας πείτε εσείς για όλα αυτά. Ευχαριστώ κύριο Σάλβαρο. Θα είμαι σύντομο. Γιατί ο Κλόντ Μωρές ήδη έθεσε τα περισσότερα ερωτήματα που ήθελα και εγώ να θέσω. Σας ευχαριστώ κύριε Γουάιν και κυρία Πρέτ που είσαστε εδώ. Μια σύντομη ερώτηση σε σχέση με αυτά που ήδη ερώτησε ο, ο Κλόντε για την Ευρωπόλ. Καταρχήν είπατε, και μάλλον το ξέρετε καλύτερα από εμά, ότι το, το έργο της Europol είναι επιβολή των, της νομοθεσίας και όχι αντικατασκοπία, η κατασκοπία. Όμως με τη συμφωνία αυτή, τη TFTP, Συμφωνείτε μαζί μου ότι η επαλήθευση του αιτήματο στον ΗΠΑ θα μπορούσε να γίνει καλύτερα από το Eurojust αντί για τη Europol. Και επίσης δεν με εκπλήσει που δεν γνωρίζετε που η NSA ή άλλες υπηρεσίες σας δίνουν στοιχεία. Μάλλον δεν θα σας το λέγανε. Σας, ε, θέλω να σας ευχαριστήσω κυρία Πρέτπε που ήρθατε για αυτές και μας ενημερώσετε. Να σας κάνω και σας μια ερώτηση. Νομίζω πως το θέμα και το καθήκον των νομοθετών είναι να υπάρχει νομική βεβαιότητα για το τι μπορεί κανείς να κάνει και τι όχι. Και ίσως η απάντηση στην ερώτηση του κυρίου Μωράς θα ήταν Μήπως υπάρχουν ε, μυστικές υπηρεσίες που έχουν βάλει πόγια καλώδια και παίρνουν τα στοιχεία από τα συστήματά σας. Ίσως εσείς να μην έχετε κάποια διαρροή, αλλά στη μεταφορά από το σημείο Α στο σημείο Β, αν κανείς ε, πάει και παίρνει στοιχεία από εκεί, ίσως να μην μπορείτε να το δείτε. Όπως σας είπα θα είμαι σύντομος και ίσως μια τελευταία ερώτηση και στους δύο. Μπορείτε να φανταστείτε σε περίπτωση που οι ισχυρισμοί αυτοί δεν ε, αρθούν τελείως, ε, μήπως ε, τελικά πρέπει να τεθεί ένα τέλος ή να ανασταλεί η ισχύ σε αυτές τις Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βος. Σας ευχαριστώ. Τέσσερις ερωτήσεις έχω να κάνω. Εσείς δεν ξέρετε αν η NSA έχει πρόσβαση στο SWIFT ή στο σύστημα δεδομένων. Υπάρχουν ε, έρευνες που να γίνονται επί τη βάση αυτών των αποκαλύψεων του τύπου και είναι δυνατόν να γνωρίζουμε από την, παρακολούθηση την παρακολούθηση συνδιαλλαγών αν αυτό έχει γίνει μέσα ε, στο σύστημα. Υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στην Europol, το SWIFT και την NSA και υπάρχουν ε, συστήματα συνεργασίας με άλλες αμερικανικές αρχές. Έπειτα, ερώτηση προς την Europol. Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις μιας ε, αναστολής του προγράμματος της ε, TFTP για την Europol και για την καταπολέμηση του, της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ, η κυρία Ιντεβέλτ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Ε, όταν ο, ο εισαγγελέας των Ηνωμένων λέει ότι πως έχετε εσείς ε, όλα τα απαραίτητα εργαλεία εντός της Europol για να διεξάγετε κυβερνού έρευνες για τα κυβερνοεγκλήματα. Εγώ όλο τυχαίως είμαι, έχω, εδρεύω στις κάτω χώρες, όπως και ο σερβερ του SWIFT. Και είδαμε ότι μας είπατε πως δεν μπορούσατε να θεσπίσετε μια εγκεκριμένη πρόσβαση στο σύστημα. Αλλά είδατε ότι αυτό το εποπτεύουν ε, θεσμοί όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα ήθελα να γνωρίζω ποιο είδο εμπειρογνωμοσύνη χρησιμοποιεί το SWIFT ώστε να, είναι βέβαι, να είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση άνευ ε, αδείας, παράνομη πρόσβαση. Μπορεί να, ε, χρησιμοποιείται κωδικούς, κρυπτογράφηση. Εγώ από τεχνικής άποψης ε, δεν ξέρω τίποτα, αλλά μάθαμε ότι ε, η Αμερικανική κυβέρνηση έχει σπάσει τα συστήματα κρυπτογράφησης και έχει βοηθήσει και οι κυβερνήσεις να παρακάμψουν τα συστήματα αυτά. Δεν με πείθει λοιπόν το επιχείρημά σας και θα ήθελα να έχω την βασική απάντηση από τον κύριο Wainwright όσον αφορά την ασφάλεια των συστημάτων. Εσείς και η μονάδα σας κυβερνοεγκλημάτων θα ερευνήσετε την ασφάλεια του συστήματος SWIFT και θα ήθελα επίσης να εκφράσω την πολύ βαθιά μου απογοήτευση και απόγνωση όσον αφορά την άρνηση του Ολλανδού Υπουργού που είναι υπεύθυνο γι' αυτό να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής μας. Γιατί λένε ναι, τα αφήνουμε σε αυτή την ομάδα εργασίας της Ένωσης και των υπαλλήλων της Ένωσης και των ΥΠΑΜΑ. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν είναι εγγυημένη ασφάλεια το σύστημά των σημαίνει αν οι μπορούν να το σπάσουν το σύστημά μας, σε οποιαδήποτε χώρα μπορεί. Πρέπει να μπορούμε να βασιζόμαστε στα συστήματά μας. Και έπειτα, το SWIFT λέει ναι, ναι, κλείνω πρόεδρε. Το SWIFT λέει ότι πρέπει να ε, ε, συμμορφωθούμε προς τα αιτήματα έρευνας άλλων χωρών. Ναι, αλλά πρέπει να συμμορφωθείτε και προς το ευρωπαϊκό νόμο πώς ε, ε, συμμορφώνεστε προς ε, τα αιτήματα έρευνας άλλων χωρών, εκτός δηλαδή των ΗΠΑ. Μάλιστα, ο κύριος Άλμπρεχτ. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για την προθυμία που επιδείξατε να έλθετε εδώ και να μιλήσετε ανοιχτά για αυτό που κάνετε. Θα ήθελα να συνεχίσω πάνω σε αυτό που ρώτησε μόλις η Σοφίντφελτ. Δηλαδή, υπάρχει αίτημα, κύριε Wainwright, από αστυνομική αρχή κάποιου κράτους μέλους να ερευνήσει μαζί με το κέντρο ε, κυβερνογκλήματος της ε, Europol, μαζί δηλαδή να ερευνήσουν ενδεχόμενες τέτοιες αυτές τις καζόμενες παραβιάσεις, διότι δεν είναι μόνο παραβίαση ασφάλειας, είναι και έγκλημα. Το κυβερνοέγκλημα είναι έγκλημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από συζητήσει ενέκρινε σχετική οδηγία. Βέβαια παράμε κάποια κρεμιστήματα, αλλά είναι προφανές και ξεκάθαρο ότι αν υπάρχει παραβίαση των συστημάτων ασφαλείας ή συστημάτων πληροφοριών στην Ευρώπη, αυτό συνιστά κυβερνό έγκλημα. Και αρχές των κρατών μελών και εσείς και το κέντρο έγκληματος θα πρέπει έπειτα να ερευνήσετε αυτά τα πιθανά εγκλήματα. Και φυσικά και οι κλιματίες δεν πρόκειται να μας βοηθήσουν στην έρευνα. Ας ρωτήσουμε λοιπόν αυτούς που ε, κάνουν κυβερνοεγκλήματα, λέτε. Μα είναι δυνατόν να, υπάρχει δυνατότητα να μας βοηθήσουν αυτοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά την νομιμότητα του αιτήματο, ερώτηση προς την κυρία Πέτρε. Λέτε ότι δεν έχετε υπόψη σας καμία μη εξωστατωμένη πρόσβαση. Ε, διερωτώ με. Τι θα πει μη εξουσιοδοτημένη. Ότι δεν την εξουσιοδοτήσατε εσείς θα πει αυτό, έτσι. Πώς αξιολογείτε εσείς αυτήν την εξουσιοδότηση ή όχι. Αν υπάρχει ένα αίτημα από την NSA βάση του προγράμματος Bull Run ή Follow the Money χωρίς ε, να εδράζεται αυτό στην ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν, δεν το εγκρίνετε, δεν το εξοδοτείτε. Φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να μιλήσετε, δεν εξοδοτείτε να μιλήσετε γι' αυτό λόγω των επιστολών που έχετε λάβει ενδεχομένω. Αλλά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Και αν δεν μπορούμε μεταξύ μας πρέπει να το αναλάβουν ε, ερευνητέ για να δουν πώς εξουσιοδοτούν οι εταιρείε τα αιτήματα. Γιατί αν εξουσιοδοτεί, εγκρίνει η SWIFT ε, αιτήματα, όχι δυνάμει του ευρωπαϊκού δικαίου, τότε θα πρέπει οι αστυνομικέ αρχές να το σταματήσουν γιατί αυτό ουσιαστικά παραβιάζει τους κανόνες περί ε, κυβερνοεγκλήματος και περί προστασίας δεδομένων θα μπορούσε να οδηγήσει σε διπλωματική αντιπαράθεση αυτό, αλλά εμείς πολιτικοί πρέπει να το επιλύσουμε πριν χρειαστεί να ξεκαθαρίσουμε άλλο τρόπο. Ähm, Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Ernst, κυρία Ράινχαρτ, κύριε Wainwright. Ε, αυτά που λέτε κάνουν σαφές ότι είναι ένα μαύρο κουτί η Ευρωπόλ και αυτό ίσως πρέπει να αλλάξει. Εγώ θα ήθελα ε, να ξέρω από εσά το εξή. Πώς βλέπετε αυτά τα, τα δημοσιεύματα που λένε ότι όλες αυτές οι πληροφορίες έρχονται από μυστικές υπηρεσίες. Πώς το εξετάζετε εσείς τεχνικά, πώς εξασφαλίζετε ως Ευρωπόλ ότι υπάρχει και ασφάλεια του συστήματος υπολογιστών σας. Πώς το κάνετε αυτό, αυτό θα ήθελα να ξέρω. Η δεύτερη μου παρατήρηση λέτε ότι δεν υπήρξε καμιά παραβίαση της συνθήκης για το SWIFT. <clears throat> δεν υπάρχει κάποια συνεργασία με την NSA, δεν υπάρχουν πληροφορίες που δίδονται στην ε, NSA, δεν υπάρχει επομένως καμία κατάχρηση της συνθήκης. Πώς ε, καταλήγεται λοιπόν αυτό το συμπέρασμα. Πώς καταλήγεται σε ένα τέτοιο πόρισμα λοιπόν. Και για την κυρία Πέτρα Λέτε ναι, ότι εφαρμόζετε τα υψηλότερα στάνταρ προστασίας των ε, δεδομένων. Είπατε ότι έχετε μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Επί ποιας βάσης το αρίεστε αυτό. Αλλά νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον αυτό που λέτε ότι δεν παίρνετε στοιχεία που προέρχονται από μυστικέ υπηρεσίε. Ποιο είναι ο μηχανισμό με τον οποίο μπορείτε να αποτρέψετε κάτι τέτοιο και να εξασφαλίσετε ότι δεν συμβαίνει. Δεν ξέρω αν είμαι κάπω αφιλή. Ίσως και άλλοι έχουν θέσει αυτό το ερώτημα, αλλά θα ήθελα να έχω μια απάντηση. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Θα έχουμε τώρα κάποιες απαντήσεις και μετά θα λάβουν το λόγο τα υπόλοιπα μέλη. Μπορείτε να απαντήσετε λοιπόν στον πρώτο γύρο. Κύριε Wainwright. Σας ευχαριστώ. Πολλά από αυτά τα ερωτήματα έχουν να κάνουν με τις σχέσεις Ευρωπόλ NSA. Δεν έχουν σχέσεις αυτοί οι δύο φορείς. Δεν έχουμε συνεργασία με αυτήν την υπηρεσία την NSA και ούτε έχουμε καμία εντολή να ελέγξουμε οποιασδήποτε υποτιθέμενες παραβιάσεις συνθήκες από αυτό το φορέμα. Δεν το, δεν το είχαμε καταλάβει αυτό, λέει ο κύριος Άλμπερτ. Κύριε Άλμπερτ, για μια ακόμα φορά, μου επιτρέπετε, η εντολή μας είναι να ελέγχουμε τα θέματα του κυβερνοεγκλήματος ετήσι των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών. Και για να απαντήσω στο ερώτημά σας, κανείς, καμία αστυνομική αρχή κράτους μέλους δεν μας ζήτησε να ερευνήσουμε <clears throat> τις, ε, τους ισχυρισμούς αυτούς και τις καταγγελίες που είναι το θέμα της έρευνάς σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσετε αυτό που προσπάθησα να κάνω σαφές ότι η εντολή της ε, Europol δεν καλύπτει τέτοιες πιθανές παραβιάσεις. Δεν καλύπτει κατασκοπία η οποία προέρχεται από εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας. Και δεν έχουμε πάρει και καμία αίτηση από κανένα κράτος μέλος για να ελέγξουμε παραδείγματος χάρη πιθανές παραβιάσεις των συστημάτων ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κίνα. Δεν είναι αυτά λοιπόν σύμμορφα με την εντολή μας. Και λόγω όλων αυτών, πραγματικά δεν ξέρουμε τι κάνει και τι δεν κάνει η NSA. <clears throat> δεν έχουμε στοιχεία στα, στους φαγγέλους μας, ακόμα και στο πλαίσιο της συμφωνίας TFTP, ώστε είτε να επιβεβαιώσουμε είτε να διαψεύσουμε αυτές τις καταγγελίες που έχουν γίνει. Δεν σημαίνει αυτό ότι η Europol δεν έχει ιδέα ή ότι ε, αποτυγχάνει στο καθήκον της. Απλώς είναι ένα άλλο κομμάτι του κόσμου με το οποίο εμείς δεν έχουμε επαφή. Δεν μας έχει ζητήσει κανείς να ερευνήσουμε περαιτέρω αυτά τα θέματα. Ο κύριος Μωράης ρώτησε και για το ρόλο της Europol στην συμφωνία TFTP και αν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Eurojust να γίνεται έλεγχος βάσει του άρθρου 4, μα αυτή ήταν μια πολιτική απόφαση που έγινε από τους νομοθέτες τότε να δοθεί αυτή η αρμοδιότητα στη Eurojust και όχι στη Europol. Μπορείτε να έχετε διαφορετική άποψη αν ήταν αυτό σωστό ή όχι, αλλά εμείς πρέπει να τηρήσουμε αυτά που αποφάσισαν οι νομοθέτες. Έχουμε συζητήσει μαζί τους όλα αυτά τα θέματα. Και σας υπενθυμίζω τις, ε, τα πρόσφατα απορίσματα σε σχέση με τη λειτουργία αυτής της διαδικασίας. Εμείς κατά τα άλλα είμαστε 100% πρόθυμοι να εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία. Αν τροποποιηθεί αυτή η συμφωνία στο μέλλον, θα πρέπει να αλλάξουμε τις διαδικασίες μας αυτή τη στιγμή είναι τεχνικού χαρακτήρα το έργο μας και έχει σαν στόχο να κάνει αυτό το οποίο μας ζήτησαν και οι νομοθέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εστιάζουμε την προσοχή μας εκεί. Ο κύριος Φως μίλησε για την ε, συμφωνία TFTP και τις επιπτώσεις της παραβίασής τους. Χρειάζεται να περιμένουμε τις θέσεις της Κομισιόν για την αξία αυτού του προγράμματος. Έχουμε συμβάλει σε αυτό το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τις ε, ε πληροφορίες που έχουμε πάρει από τις Ηνωμένες Πολιτείες χάρη στο TFTP. Αλλά αυτό δεν είναι στα τρέχοντα που μας ενδιαφέρουν σήμερα. Και ένα ακόμα σημείο. Αυτό που είπε η κυρία, αυτό που ρώτησε η κυρία Ένστ για την ασφάλεια των πληροφορικών συστημάτων της Europol. Λόγω της εντολής μας, ως κέντρο κυβερνο, αντιμετώπισης κυβερνο εγκλήματος. Τα παίρνουμε αυτό πάρα πολύ στα σοβαρά. Και λόγω της υποχρέωσής μας να προστατεύουμε προσωπικά δεδομένα, η Europol έχει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε κάποια αστοχία στα συστήματα ασφάλειάς μας, χάρη στα επενδύσεις που κάναμε να είναι όσο δυνατόν πιο ανθεκτικό αυτό το σύστημα. Αυτά νομίζω για τον πρώτο γύρο. Η ε, κυρία Πέτρο, σας ευχαριστώ. Και εγώ θα απαντήσω στο πρώτο ερώτημα για τη διακίνηση δεδομένων βάσει τη SWIFT. Κλείνει το μικρόφωνο της ομιλήτρια. Um, Μπορεί να μην ξέρουμε, αλλά είναι δυνατό οι τράπεζες που στέλνουν δεδομένα μέσω της SWIFT μπορούν να τυπώσουν αυτά τα μηνύματα και μετά να κάνουν διακίνηση αυτών των δεδομένων μέσα στο εσωτερικό του σύστημα και ίσως η NSA έχει μπορέσει να διαβάσει αυτά τα τυπωμένα μηνύματα. Αυτή είναι η εξήγηση που δίνουμε. Και πώς ξέρουμε ότι δεν μας παρακολουθούν, τι πρότυπα χρησιμοποιούμε, τι κρυπτογράφηση χρησιμοποιούμε είναι δύσκολο να αποδείξει κανείς ότι δεν σε παρακολουθούν. Αυτό που προσπάθησα να εξηγήσω είναι ότι έχουμε πολλά συστήματα ελέγχου της ασφάλειας για να εντοπίσουμε τις ε, μη νόμιμες προσπάθειες πρόσβασης για την κρυπτογράφηση. Τα υψηλότερα διεθνή ε, πρότυπα για το μηχανισμό μας ε, κρυπτογράφησης και χτες ο κρυπτογράφηση κρυπτογράφησης της SWIFT μου είπε ότι τα συστήματα αυτά τα έχουν επινοήσει οι δύο Βέλγοι. Ξεκίνησαν από την Ευρώπη. Και μου είπε αυτός ο εμπειρογνώμων ότι χρησιμοποιούμε εμπειρογνώμονες τρίτων φορέων. <clears throat> Συνεργαζόμαστε με πανεπιστήμια, με ιδιωτικούς εμπειρογνώμονες ασφάλειας και λειτουργούμε εδώ με το Πανεπιστήμιο του Λουβέν στο Βέλιο. Τώρα, ποιος έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Τα στοιχεία που έχουμε είναι τα στοιχεία των πελατών μας. Οι πελάτες μας λοιπόν μπορούν να <clears throat> έχουν πρόσβαση. Και εμείς πάντα λέμε στους πελάτες μας ότι δεν θα δώσουμε ποτέ εθελοντικά τα στοιχεία τους σε κάποιο τρίτο φορέα. Αυτό είναι μια βασική αρχή. Πρέπει να έχουμε να μας υποχρεώσουν σε νομικό επίπεδο να πάρουμε μια νομικά δεσμευτική αίτηση, να δώσουμε στοιχεία σε μια αρχή για να τα δώσουμε. Είμαστε μια παγκόσμια εταιρεία βέβαια και πολλοί φορές μπορούμε να βρεθούμε μέσα σε δύο διαφορετικά νομικά συστήματα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο θα δημιουργήσει ασφάλεια δικαίου για να επιτρέψουμε στη SWIFT να λειτουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Νομίζω πάρεις να απαντήσω. Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να έχω ε, γραπτή απάντηση στις ερωτήσεις που κάναμε στην εταιρεία SWIFT να τις λάβουν γραπτός και να μας απαντήσουν γραπτός. Δεν απάντησε τίποτα εκπρόσωπος. Επίσης, κύριε Winwright κανένα κράτος μέλος δεν ζήτησε από την Ευρωπόλ να ερευνήσει ενδεχόμενη ε, παραβίαση ή δυνατότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ε, στο διακομιστή. Κανένας δεν ζήτησε έρευνα. Και αν είναι αλήθεια αυτό δεν είναι αξιοπερίεργο. Πρόεδρος, πριν σας ξαναδώσω το λόγο θα έλεγα να ακούσουμε πρώτα τους άλλους βουλευτές. Ε, ε, ή μήπως θέλετε εσείς να απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Ναι, ορίστε. Σωστά ε, τα είπατε κύριε τα δεν λάβαμε έτοιμα από κανένα κράτο μέλο να ερευνήσουμε οποιαδήποτε καζόμενη παραβίαση σε σχέση με οποιαδήποτε πτυχή τη έρευνα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς η Επιτροπή σας, δηλαδή, ούτε και σε ό,τι αφορά μια εξουσιοδοτημένη διείσδυση στο SWIFT. Let's, let's open some floor for the rest of the members. I suggest... Να δώσω τώρα το λόγο σε όποιον άλλο βουλευτή θέλει το λόγο, αλλά πάλι ε, δύο λεπτά το πολύ, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και έχουμε πολλούς βουλευτές. Πίρκερ. Σας ευχαριστώ. Εγώ χαίρομαι για το γεγονός ότι από τον κύριο Wainwright και την κυρία Πέτρα υπήρξαν κάποιες διευκρινήσεις. Υπάρχουν τόσες πολλές υποψίες και κατηγορίες που κυκλοφορούν ώστε νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε σαφήνεια σε σχέση με το ρόλο της Europol. Είναι μια, ένας φορέας ε, εφαρμογής του νόμου και όχι ένας φορέας αντιμετώπισης της κατασκοπίας. Είναι καλό λοιπόν ότι όλα αυτά που κάνει η Europol γίνονται κάτω από νομικό έλεγχο. Αναφέρατε επίσης κύριε Wainwright ότι έχετε μια πολύ καλή συνεργασία με τις ποινικές με τις διοκτικές αρχές για ποινικά αδικήματα στις ΗΠΑ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω με ποιες αρχές των ΗΠΑ έχετε συνεργασία σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του εγκλήματος. Μήπως μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα και μήπως μπορείτε να μας πείτε σε ποιους βαθμούς, σε ποια σημεία ήταν καρποφόρα αυτή η συνεργασία και οδήγησε σε θετικά στοιχεία και επίσης προς την κυρία Πέτρε. Θα ήθελα να πω, έχετε κάποιες ενδείξεις ότι στοιχεία τα οποία προήλθαν από το δικό σας σύστημα έχουν μεταδοθεί σε αρχές οι οποίες δεν είχαν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε αυτά μέσω της παρέμβασης ε, άλλων φορέων. Κυρία Ζίπελ, θέλω να μην επαναλάβω αυτά που είπαν <clears throat> οι άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ την κυρία Πέτρα γιατί κάνετε σαφές με σε πόσους χώρους και με ποια, σε ποια επίπεδα γίνεται η προστασία των δεδομένων. Θα ήθελα όμως να θέσω το ερώτημα στην Europol αν έχετε και εσείς αντίστοιχες διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων και μπορείτε να πείτε το ίδιο και με τη SWIFT. Μπορεί να υπάρξει η δυνατότητα μια εταιρεία να δώσει σε μια άλλη εταιρεία τις κλίδες για τα δικά της πληροφορικά προγράμματα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίσω εγώ είναι ότι κανείς δεν μπορεί να ελέγχει αν πράγματι τα πράγματα λειτουργούν όπως λέγεται ότι λειτουργούν. Λέτε ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών παίρνει μονάχα αυτά τα οποία τους δίνουμε εμείς, αλλά κανείς δεν εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει συλλογή δεδομένων με άλλο τρόπο. Και ένα τελευταίο ερώτημα, όχι για σήμερα, αλλά το οποίο πρέπει να συμβάλλει στην μελλοντική συζήτηση. Αν δεν είναι αρμόδια η Europol για να αντιμετωπίσει παραβιάσεις ε, προσωπικών δεδομένων στη SWIFT σε άλλες βάσεις δεδομένων. Όταν πρόκειται για παραβίαση που προέρχεται από μια κρατική αρχή. Ποια ευρωπαϊκή αρχή είναι αρμόδια για να μας προστατεύσει και πώς συντονίζονται οι εθνικές αρχές και τι γίνεται αν μια εθνική αρχή δεν δέχεται να συμμετάσχει σε αυτή την προστασία. Κυρία Λάτφορντ. Σας ευχαριστώ. <clears throat> Το ίδιο ερώτημα ε, ισχύει και όπως και για τις τηλεφωνικές εταιρείες και τις εταιρείες παροχής ε, υπηρεσιών ίντερνετ. Για μένα όλα αυτά καταλήγουν στο ερώτημα του κατά πόσο τα συστήματα που αποτελούν τον πυρήνα του SWIFT είναι υπονομευμένα ή αν υπήρξε κάποια συγκατάβαση, συγκατάθεση στις ε, αιτήσει της NSA από την πλευρά της SWIFT. Να είμαι σαφής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα μου πείτε, δεν θα απαντήσω. Συνεργάζεται η SWIFT με αιτήσει, με δικαστικές κλητεύσεις ή οποιαδήποτε άλλη αίτηση να δώσει στοιχεία πέραν του πλαισίου της ε, συμφωνίας TFTP. Γιατί ρώτησε η Σοφή τι κάνει η SWIFT με δικαστικές κλητεύσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι κάνει όμως με κλητεύσεις μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέτε ότι γίνεται αυτό μόνο μέσα στα πλαίσια του TFTP. Ε, μήπως γίνεται και εκτός αυτού. Και επίσης χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θα σας πληροφορούσαν αν έχουν πάρει μια κλήτευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από κάποιον άλλο. Πόσο μεγάλη εποπτεία έχετε λοιπόν για όλα αυτά τα θέματα. Εγώ βλέπω ότι αυτές οι καταγγελίες ήταν πραγματικά σοκαριστικές για το γεγονός ότι έχουν υπονομευθεί και τα συστήματα κωδικοποίησης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση όλης της παγκόσμιας οικονομίας και το SWIFT, το σύστημα SWIFT είναι κεφαλαιόδες για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των συναλλαγών στο διαδίκτυο. Όλα αυτά λοιπόν που έχουν να κάνουν με την επιγραμμική οικονομία, της συναλλαγής στο διαδίκτυο, έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη. Αν, υπάρχει, αν υπάρχουν στα προγράμματα αυτά λοιπόν οι θελημένες παρα, οι θελημένες τρύπες και παραθυράκια, αυτό είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και πράγματι θα ήθελα να ξέρω ποιο ερευνά όλα αυτά τα θέματα. Δεν βλέπω κάποιον είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, είτε εδώ στι Βρυξέλλε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να λέει ότι εγώ τα ψάχνω αυτά τα θέματα και προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Μα είναι κάτι που μας αφήνει εμβρόντιτους. Κύριε Wainwright, εσείς υποτίθετε ότι είσαστε επικεφαλής του, της Ευρωπαϊκής Μονάδας για το έγκλημα. Τι νόημα έχει να μιλάμε για κυβερνό έγκλημα και να μην κάνετε τίποτα. Ο επικεφαλής της ε, ε, του προσωπικού της υπηρεσίας μου έδωσε κάποιες επαφές στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί αλλιώς δεν μπορούσα να βρω κανέναν στο Ηνωμένο Βασίλειο που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Τουλάχιστον μου έδωσε κάποια, ε, κάποιο σημείο επαφή στη Βρετανική αστυνομία γύρω πόλ. Κυρία Μορβάη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω κι εγώ να μιλήσω εξ ονόματος των Ευρωπαίων πολιτών και των Ούγκρων πολιτών και να πω ότι πρέπει τα πράγματα να ξεκαθαριστούν. τα εμπιστευτικά τραπεζικά δεδομένα, απόλυτα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών, με τον ένα τον άλλο τρόπο βλέπουμε ότι μπορούν να αποκτηθούν από τις ε, αρχές των ΗΠΑ. Έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Αυτές ε, οι υπηρεσίες, ε, μυστικές κτλ. έχουν δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών στη διάθεσή τους και υπάρχουν, ε, ε, υπάρχει αυτή η διμερή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα που ρυθμίζει, ρυθμίζει την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Αυτή είναι η αρχή όμως. Μήπως ξεπερνούν το πλαίσιο αυτής της συμφωνίας των Πολιτείες και πηγαίνουν πιο πέρα. Ο πατριωτικός νόμος δίνει στις ΙΠΑ τη δυνατότητα να απαιτήσουν, όχι απλά να αιτηθούν, αλλά και να απαιτήσουν ε, τραπεζικά στοιχεία ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Αν δει κανεί ε, την ομολογία και τα σχετικά με τη βίζα, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο επίπεδα πρόσβασης στις πληροφορίες. Δηλαδή επιβάλλονται δύο επιπέδων απαιτήσει, αν θέλετε. Έχουμε από τη μία πλευρά τις γενικές διαδικασίες ποινική ε, ε, ε, παραβίασης. Και έπειτα υπάρχει και ένα δεύτερο σύστημα εγγυήσεων σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία. Είναι ένα σύστημα εγγύησης ασφαλιστικής δικλίδας, δεν ξέρω καν πώς να το πω θα έλεγα ότι πάει πολύ πιο πέρα. Άγρα πληροφοριών επιτρέπεται χωρίς κανένα όριο. Μιλάμε εδώ για δραστηριότητες, για ενέργειες που συνιστούν παραβίαση του ποινικού δικαίου. Έχουμε την Ευρωπόλ, έχουμε από την άλλη πλευρά όμως την Αμερικανική κυβέρνηση και έχουμε και το Υπουργείο Οικονομικών τέτοιο ε, είναι αυτό το, το πλαίσιο το οποίο εμείς θέλουμε να ισχύει και αυτό το, σε αυτό συμφωνούν και οι Ηνωμένε Πολιτείες. Όπου θέλουν, είπα, ισχύει ο πατριωτικός νόμος. και το σύστημα εγγύησεων ε, που ισχύει θα είναι πολύ λιγότερο αυστηρό ώστε να μπορούν είπα να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες. Πρέπει επίσης να ενημερώνονται οι πολίτες. Σε πόσες περιπτώσεις ε, δόθηκαν πληροφορίες, ε, ενημερώθηκε ο πολίτης για τον, τα οποία του οποίου τα στοιχεία δόθηκαν ή τα απέκτησαν οι νόμες πολιτείες. Ρομέρο. Προς τον κύριο μια ερώτηση που είπε ότι η Ευρωπόλ ναι, είναι μια πολιτική απόφαση. Πράγματι γνωρίζουμε ότι είναι ένα αστυνομικό όργανο το οποίο έχει αναλάβει και την προστασία δεδομένων. Βέβαια, αυτά τα δύο θα μπορούσαν και σήμερα μεταξύ του ε, ω καθήκοντα του ίδιου οργάνου. Αλλά εμεί θα πρέπει αυτό να το αναλύσουμε στο μέλλον για να δούμε πώ ε, θα μπορούσαμε να πετύχουμε ε, να έχουμε ένα μια σωστή διαδικασία. Σε ό,τι αφορά αυτή όμω τη συμφωνία τη FTP. Εδώ δεν μιλάμε για, για αυτή τη συμφωνία και για τις παρακολουθήσεις ή διαρροές που υπήρξαν. Έχετε πληροφορίες ότι υπήρξαν ή όχι. Και τι συνέχεια δόθηκε. Και σε ό,τι αφορά την κυρία Πέτρε. Αυτό το μνημόνιο, αυτή η συμφωνία με τη ΣΥΠΑ που έχετε με τη ΣΥΠΑ για να τους δίνετε πληροφορίες. Δίνετε κρυπτογραφημένες πληροφορίες. Δεν τους δίνετε και κάποιο κλειδί, γιατί αλλιώς γιατί τους τα στέλνετε κρυπτογραφημένα, Γιατί νόημα έχει τι ε, πληροφορίες υποχρεούστε να δώσετε και υπό ποιους όρους έχετε ε, στοιχεία να μας δώσετε. Αυτό το μνημόνιο τι λέει, τι προβλέπει. Υπάρχει επίσης αυτές 200 χώρες στις οποίες ε, ασκείται δραστηριότητα. Υπάρχει κάποιες φορές που σας ζήτησε αντίστοιχες πληροφορίες με αυτές που σας ζητήθηκαν από τις ΗΠΑ ή υπάρχει κάποια συμφωνία, σύμβαση, σύμφωνο με κάποιο άλλο κράτος εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχετε υπογράψει και έχετε υποχρέωση να δίνετε και σε αυτούς τέτοιες ε, πληροφορίες. Ευχαριστώ. Thank you. the last intervention, Mr. Bronze. Κύριος Μπρόντς, ο τελευταίος που θα το λόγο. <clears throat> Σας ευχαριστώ. Μας διαβεβαίωσε η Europol ότι δεν έχει καμία σχέση με την ε, NSA ή τη CIA στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχει καμία σχέση και με τις υπηρεσίες ασφαλείας των κρατών μελών δεν παίρνει πληροφορίες από αυτές. Τα στοιχεία που κρατάει η Europol περιορίζονται σε άτομα που είναι ύποπτοι εγκλημάτων. Θα μπορούσε να είναι ευρύτερα τα στοιχεία αυτά και για άτομα τα οποία δεν είναι ύποπτοι εγκλημάτων γιατί η αστυνομία του Λονδίνου χρησιμοποιεί την ίδια διοικητική ομάδα για να αντιμετωπίσει και την βία πολιτική δράση και την τρομοκρατία από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά τα άτομα τα οποία είναι εξτρεμιστές σε πολιτικό επίπεδο. Για το κυβερνό έγκλημα. Ακούσαμε να μας λέτε ότι η Ευρωπόλ έχει την υποχρέωση να ε, ερευνά το κυβερνό έγκλημα αιτήσει των κρατών μελών, αλλά δεν έχει πάρει καμία τέτοια αίτηση μέχρι στιγμής. Μήπως έχει την ευθύνη να ερευνά καταγγελίες από άτομα και Φόρης εναντίον των κρατών μελών ή εναντίον κυβέρνησεων τρίτων χωρών εάν υπήρχε η υποψία ότι κάνουν εγκλήματα στο διαδίκτυο. Κυρία Πέτρα, <clears throat> είπατε ότι έχει μηδενική ανοχή το SWIFT σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις προσωπικής ασφάλειας. Μήπως ε, κάποια μέλη του προσωπικού έχουν κάνει μια τέ, τέτοιες παραβιάσεις της ασφάλειας και πώς τους αντιμετωπίσανε. Μας είπατε ότι δεν υπάρχουν καθόλου παραβιάσεις από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Έχουν δείξει οι <clears throat> έρευνες σας κάποια προσπάθεια παρίσφρησης στα δεδομένα από μυστικές υπηρεσίες ή από κάποιους που είναι ύποπτοι να εργάζονται με μυστικές υπηρεσίες. Και είπατε επίσης κύριε Πέτρε ότι αν σας υποχρεώσουν να δώσετε δεδομένα θα πείτε και στους εμπλεκόμενους μήπως οι νόμοι κάποιας χώρας θα την εμπόδιζαν να κάνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Ιντφέλτ για μια σύντομη παρέμβαση. Ναι, ζητώ συγγνώμη στους συναδέλφους που ξαναπαίρνω το λόγο, αλλά κάποιος μου τόνισε και διορθώστε με αν κάνω λάθος, πως η ίδια η Ευρωπόλ θα είχε το δικαίωμα να ζητήσει από τα κρατημέλη να ξεκινήσουν μια έρευνα για διεθνή εγκλήματα. Είναι, δυνατόν λοιπόν τεχνικά και θεωρητικά η, ε, Europol ε, να ζητήσει από ένα κράτος μέλος, ας πούμε την Ολλανδία, να διεξάγει σχετική έρευνα για αυτή την υπόθεση. Ο κύριος Βάινραιτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σπίρκε ρώτησε τι συνεργασία έχουμε με τη ΣΥΠΑ. Δεν θα μακρηγορήσω. Έχουμε πάρα πολλές ε, συνεργασίες σε κάθε τομέα του διεθνούς εγκλήματος, με το FBI, με την ε, ε, υπηρεσία αντιμετώπισης των ναρκωτικών κτλ. Πολλά γίνονται και στον τομέα τον ε, του κυβερνοεγκλήματος και έτσι έρχομαι στην απάντηση προς τη Σάρα Λάτφορντ εφόσον δεν το κάνουμε αυτό γιατί δεν κάνουμε κάτι άλλο. Είμαστε πάρα πολύ απασχολημένοι. Έχουμε ένα πολύ μακρύ κατάλογο δραστηριοτήτων για το έγκλημα που περιλαμβάνουν για παράδειγμα την κατάχρηση των των ανθρώπων, της, την, την κατάχρηση δισεκατομμυρίων ε, ευρώ online ε, και όλα αυτά με τις μη εγκεκριμένε δραστηριότητες ε, εγκληματικών οργανώσεων στο ίντερνετ. Δεν έχουμε συγκεκριμένους ισχυρισμού για παράνομες δραστηριότητες από κυβερνήσεις. Δεν είναι κομμάτι της εντολής μας αυτό. Και παράλληλα, σε σχέση με αυτό το θέμα για την κωδικοποίηση, την κρυπτογράφηση που αναφέρατε κύριε Λάτφορτ, Εμείς στη Europol θεωρούμε πως τα στάνταρ ε, της ε, κρυπτογράφησης είναι αρκετά απαιτητικά και η εξαγωγή ή ε, ε, ε, το, το σπάσιμο τέτοιων κρυπτογραφημένων πληροφοριών είναι μεγάλη δυνατότητα για τις εγκληματικές οργανώσεις Τελευταία μάλιστα είχαμε μια μεγάλη, ένα μεγάλο επίτευγμα όσον αφορά την κατάχρηση παιδιών ή την κακομεταχείριση παιδιών. Προσπαθούμε και να έχουμε όσο γίνεται πιο ψηλά στάνταρ κρυπτογράφησης που να μην μπορεί κανείς να τα σπάσει και αυτό δίνει την ευκαιρία να μην δίνουμε ευκαιρία μάλλον στους εγκληματίες. Είναι μια συνέπεια την οποία θα πρέπει να γνωρίζουμε. Καμιά φορά είναι πάρα πολύ δύσκολα να αποκρυπτογραφηθούν όλα αυτά. Τώρα, για την ερώτηση Ρομέρο Λόπες. Δεν έχουμε αποδείξεις ε, για παραβίαση της συμφωνίας TFTP από πλευρά των ΗΠΑ και επαναλαμβάνω απλά αυτά που είπε η κυρία Μάλστρομ προηγουμένω. Από τη δική μα εμπειρία, οι ΗΠΑ ε, δεσμεύονται και εφαρμόζουν ε, όλε τι συμφωνίε και όλα όσα αφορούν την Europol και μάλιστα βελτιώνεται η συνεργασία μας ε, ε, κατά τη διάρκεια των τριών ετών εφαρμογής της ε, συμφωνίας. Γιατί όσο είπε ο κ. Μπρόνζ, δεν έχουμε άμεση συνεργασία με την CIA ή την NSA. Έχουμε παραδοσιακά συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφαλείας των κρατών μελών. Είμαι συγκεκριμένα μέλη οι εντολές που μας δίνει το Συμβούλιο για τα καταπολέμηση το, της τρομοκρατίας. Όμως ε, αυτό γίνεται σποραδικά και δεν είναι σημαντικό σε σχέση με την φύση γενικότερα των εργασιών μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10-15 ετών. Τώρα, από ποιον παίρνουμε ε, στοιχεία. Αυτό ε, προβλέπεται εξ αρχής για τους φακέλους που έχουμε στην Europol και καθένας από τους φακέλους ευκρινίζεται πολύ συγκεκριμένα η φύση της ποινική δραστηριότητας για την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα. Θα δείτε λοιπόν πως υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι ορισμοί, αυστήρα ελέγχονται από τις αρχές προστασίας των δεδομένων για συγκεκριμένους τύπους εγκλημάτων όπως ας πούμε η εμπορία ηρωίνης, ορισμένες μορφές κυβερνό εγκλημάτων κτλ. Ε, δεν έχουμε δυνατότητα να ερευνήσουμε κυβερνήσεις. Ε, η κυρία Ίντφελτ ε, είπε κάτι σωστό. Είναι αλήθεια ότι στο νομικό μας πλαίσιο υπάρχει δυνατότητα η Europol να ζητήσει από κάποιο κράτος να ερευνήσει ύποπτες, υποψίες για εγκληματική δραστηριότητα με την έννοια ότι βέβαια που εντάσσεται στην εντολή μας. Δεν επεκτείνεται όμως στις κρατικές δραστηριότητες η εντολή μας και γι' αυτό νομίζω θα είχαμε μια νομική ε, δυσκολία να υποβάλουμε τέτοιο αίτημα. Πάντως, δεν, έχω, δεν είμαι απόλυτα ενήμερος για να σας απαντήσω, για να είμαι ειλικρινής. Πάντως είναι καλό το ερώτημά σας. Ευχαριστούμε. Η κυρία Πέτρε. Σας ευχαριστώ. Για το ερώτημα του πώς γνωρίζουμε ότι τα στοιχεία δεν δίνονται σε μη εγκεκριμένου εταίρου. να προσθέσω κάτι σε σχέση με αυτό που είπαμε πριν. Καταρχήν η συμφωνία TFTP ε, αναφέρεται σε μετέπειτα μεταφορά. Δηλαδή, τα στοιχεία που παίρνει κανείς από το TFTP να μπορούν να δοθούν σε άλλες αρχές. Δεύτερον, ε, αυτό που θέλω να πω είναι και πάλι ανησυχία για το SWIFT, όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί και προσπαθούμε να έχουμε σαφήνεια για όλα αυτά. για το θέμα του προγράμματος και την πρόσβαση άλλων αρχών, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι το μόνο πρόγραμμα που υπάρχει και δεν έχουμε παρόμοια προγράμματα στον υπόλοιπο κόσμο αν εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ε, να ανταποκριθούμε σε κλητεύσεις. Ε, ναι, βεβαίως ε, από καιρούς καιρών θα πρέπει να συμμορφωνόμαστε με νομικά δεσμευτικές κλητεύσεις. Υπήρχε ακόμα ένα ερώτημα. Γνωρίζουμε εάν οι τράπεζες ή πότε οι τράπεζες υπόκεινται οι ίδιες σε κλητεύσεις όταν λαμβάνουν τέτοιου είδους ε, δεσμεύσει, μάλλον ανακοινώσει και δεν, ξέρω και δεν ξέρουμε πόσε λαμβάνουν οι τράπεζε, πόσε ε, πόσες κλητεύσεις και ούτω ή άλλω είναι υποχρεωμένε να αναφέρονται στις εποπτικές του αρχές και να αναφέρουν τι πληροφορίες για τους πελάτες ή για εγκληματικές υποθέσεις. Υπήρξε και άλλη μια ερώτηση Αν υπήρξαν περιπτώσεις που μας εμπόδισε ο νόμος να ενημερώσουμε τους πελάτες μας. Ε, μα ε, οποιοδήποτε ζητείτε να δώσει πληροφορίες θα πρέπει να είναι εχέμηθος σχετικά με αυτές. Δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο και πάλι αν μας υποχρεώνει ο νόμος να μην αποκαλύψουμε στον πελάτη μας ότι έγινε σχετικό αίτημα, δεν θα το αποκαλύψουμε βεβαίως. Η κρυπτογράφηση ε, Πολύ πρακτικές ερωτήσεις ε, τέθηκαν. Ε, τι κάνουμε δηλαδή όταν ε, δίνουμε τα στοιχεία που ζητούνται με τη συμφωνία TFTP. Αυτό που κάνουμε είναι αποκρυπτογραφούμε τα στοιχεία και τα δίνουμε αποκρυπτογραφημένα στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν θα τους δώσουμε κρυπτογραφημένα στοιχεία. I think I've responded to, to all the questions if I... Νομίζω πως απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Σας ευχαριστούμε κυρία Πέτρε. κυρία Λάτφορτ ζήτησε το λόγο. Σύντομα, αν μου επιτρέπετε να επανέλθω στον κύριο Βάιν Ράιτ. Ίσως να μην ε, ήμουν σαφής. Εγώ δεν διαμαρτύρομαι. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι οι εγκληματίες μπορούν να εκμεταλλευθούν και ακόμα και τις πιο σίγουρες προδιαγραφές κρυπτογράφησης. Τα κράτη φυσικά θέλουν να έχουν όσο γίνεται ψηλότερε προδιαγραφέ κρυπτογράφηση. Εμεί διαβάζουμε όμω ισχυρισμού ότι μπορεί να μην του ενδιαφέρει αυτό. Να μην έχουν δηλαδή ε, χρησιμοποιήσει τα πιο εξελιγμένα στάνταρ ε, κρυπτογράφηση και υπηρεσίες ε, αντικατασκοπίας φαίνεται να ενδιαφέρονται και να έχουν συμφέρον να υποβαθμίζουν τις προδιαγραφές κρυπτογράφηση. Εγώ θέλω να ξέρω ποιος στο επίπεδο της πολιτικής και εσείς καταστήσατε σαφές πως η δική σας εντολή δεν σας επιτρέπει να μπαίνετε στα χωράφια τη κρατική κατασκοπία. Αλλά σίγουρα η αστυνομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όλες οι εταιρείε που είναι online πάει να πει ότι μπορεί ο καθένα να μπαίνει και να κάνει ό,τι θέλει. Μα πρέπει να γίνει κάποια δημόσια συζήτηση. Και με βλέπετε κάπω ταραγμένη, αλλά όντω ε, είμαι ταραγμένη. Τι, τι είδου προστασία. Δεν το πιστεύω δηλαδή ότι είμαστε τόσο απροστάτευτοι. Πρέπει να δώσω το λόγο στην κυρία Μορβάη, αλλά μόνο για ένα λεπτό. Και μετά κλείνουμε. Ευχαριστώ. Δεν πήρα καμία απάντηση σε κανένα από τα ερωτήματά μου ρωτώ τον εκπρόσωπο της Europol αν επιτρέπεται ή αν είναι δυνατόν ότι έχουν τη δυνατότητα με τις δικές τους νομικές βάσεις να συλλέγουν στοιχεία από τους ε, Ευρωπαίων πέραν της TFTP και από την εκπρόσωπο της SWIFT. Θα ήθελα να τη ρωτήσω πόσες αιτήσει είχατε για δεδομένα που αφορούν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης <clears throat> επί τη βάση είτε λόγω τη συμφωνίας για την καταπολέμηση χρηματοδότησης τη τρομοκρατία ή γενικά από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, please, Mr. Wainwright. Κύριε Wainwright, συγγνώμη που δεν απάντησα το ερώτημά σας. Δεν ξέρω αρκετά για το νομοθέτημα Patriots ώστε να ξέρω αν ήρθανε κάποιες αιτήσει μέσω του Patriot Act για τη Europol. Ξέρω ότι οι Αμερικανικές αρχές οι οποίες καταπολεμούν την τρομοκρατία θα χρησιμοποιούν όλο το πλωστάσιο <clears throat> νομικών εργαλείων που περιλαμβάνουν και νομικές αποφάσεις και κλητεύσεις. Νομίζω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έκαναν σαφέ επίση ότι το κάνουν αυτό εδώ και πολλά χρόνια, όπω το κάνουν όλε οι χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω αρκετά όμω για το νομοθέτημα Patriot για να σα απαντήσω. Η κυρία Πέτρε, πόσε αιτήσει έχουμε πάρει <clears throat> βάσει τη συμφωνία TFTP, δεν ξέρω απ' έξω, αλλά νομίζω ότι υπήρξε μια έκθεση που δίνει κάποιον αριθμό. Αν έχουμε πολλές κλητεύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή όχι, όχι, όχι. Και αν δείτε αυτές τις ε, κλητεύσεις, οι περισσότερες απορρίπτονται γιατί δεν είναι σύνομες ή γιατί δεν ξέρουμε. Νομίζουν όλοι ότι τα ξέρουμε όλα ότι έχουμε στοιχεία πελατών. Όχι, έχουμε απλώς μηνύματα από τη μια τράπεζα στην άλλη. Η απάντηση λοιπόν είναι όχι. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μωράης θα συμπεράνει το απόγευμα από ό,τι κατάλαβα και όχι τώρα όταν τελειώσει όλη η σειρά των συναντήσεων γιατί τώρα θα, συνεχίσουμε στις 3. Σας ευχαριστώ λοιπόν συνάδελφοι για την ενεργή σας συνεργασία και ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας για τις πληροφορίες που μας έχουν δώσει. Και θα συνεχίσουμε την έρευνά μας στις 3. Τώρα πηγαίνουμε στην κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.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 περνάμε στην ε, κανονική ημερήσια διάταξη της ε, ΛΥΜΠΕ. όπου έχουμε να εξετάσουμε την ε, μεσοπρόθεσμη έκθεση για την συνθήκη αυτή, ε, καταρχήν να συγκρίνουμε την ημερήσια διαταξία. δεν υπάρχουν αντιρρήσει, ε, θεωρούμε ότι συμφωνείτε όλοι, δεν υπάρχουν ανακοινώσει, άλλε. Και απλώς ε, να εγκρίνουμε τη, τα πρακτικά τη τελευταία μα συνεδρίασης, του 9 Ιουλίου δηλαδή, 2013. Εγκρίνονται λοιπόν και έτσι προχωράμε στο σημείο 4 για την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος τη Στοχόλμη. Κοινή συνεδρίαση. Λίμπε Αύκο Γιούρι. Για να μιλήσουμε για το, την αξιολόγηση του προγράμματος. Σήμερα είχαμε κάνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και πριν το καλοκαιρινέ διακοπές και τώρα θα εξετάσουμε τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους συνεισηγητές. Είμαι και εγώ ίδιος συνεισηγητής για την ε, ΛΥΜΠΕ, αλλά θα ακούσουμε πρώτα τους συνεισηγητές από την Γιούρη και την Νάφκο. τον κύριο Μπερλιγκουέρ και τον κύριο Καζίνη. Και μετά θα κάνουμε, θα κάνουμε κάποια σχόλια σε σχέση λοιπόν με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Ας, συνεχίσουμε, ας ξεκινήσουμε μάλλον με τους συνεισηγητές. Και εγώ θα κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Ποιο θα ήθελε να ξεκινήσει, ο κύριο Μπερλιγκουέρ ή ο κύριο Καζίνη. Ο κύριος Μπερλιγκουέρ, που είναι εισηγητής για την ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια σωστή πρωτοβουλία την προώθηση της ενδιάμεσης αναθεώρησης του προγράμματος Στοκχόλμης από τις επιτροπές της Και αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο από τα έγγραφα που έχουμε υποβάλει εμείς ως συζητητές, αλλά και από τον πλούτο των τροπολογιών που υπευλήθησαν για τη συνέχιση της συζήτησης. Εγώ θα σταθώ μόνο σε κάποιους γενικούς προβληματισμούς ως προς το θέμα. Καταρχήν, μια σειρά τροπολογιών αφορά την ανάγκη να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών και άρα την ε, κατασκευή του Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης. Και γι' αυτό κάποιες από αυτές τις τροπολογίες υποδεικνύουν το, τον τρόπο μείωσης των νομικών ε, φραγμών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στη στιγμή της άσκησης του δικαιώματος της ελευθερίας κυκλοφορίας, ούτως ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στην Επιτροπή Γιούρη αναπτύσσεται μία συζήτηση ένας προβληματισμός για το πρόβλημα της αυτόματης και εύκολης αναγνώρισης ε, των ε, εγγράφων οικογενειακής κατάστασης ε, για τους πολίτες. Δεν είναι λίγο αυτό, γιατί τα έγγραφα, τα πιστοποιητικά τα διαφόρων ειδών φαίνεται κάτι light σε σχέση με τα μεγάλα θέματα της δικαιοσύνης. Δεν είναι όμως αλήθεια. Ένας Ευρωπαίος πολίτης πρέπει να αισθάνεται Ευρωπαίος πολίτης πάντοτε και δεν πρέπει διαρκώς να πρέπει να αποδείξει ότι τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του είναι τα κρατικά έγγραφα, ας πούμε, τα, πτυχία, ε, την άσκηση επαγγέλματο, την ταυτότητά του. Διαρκώς να πρέπει ξανά και ξανά να τα αποδεικνύει. Λοιπόν, τα έγγραφα, λοιπόν, ε, όπως είπαμε, ε, τα κρατικά να μπορούν να ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια και τα δικαιώματά του σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν κατατεθεί σχετικές τροπολογίες. Εν γέννη φαίνεται να είμαστε υπέρ της ενίσχυσης της νομικής κουλτούρας, της ευρωπαϊκής νομικής κουλτούρας, ιδιαίτερα για τους πτυχές εκεί όπου θεωρούμε το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι δικό μας όλων. Είναι οι αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της αρχής της επικουρικότητας, της ανεξαρτησίας της εισαγγελίας και όλη αποδοχή και όχι μόνο μερική αποδοχή του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και αυτός είναι ένας τρόπος να είναι κανείς Ευρωπαίος και είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη και την εξέλιξη μάλλον της κατάστασης. Υπογραμμίζεται η αναγνώριση της διαφοράς των άλλων ε, νομικών συστημάτων από το ένα κράτος στο άλλο και άρα αμοιβαία εμπιστοσύνη στην ποιότητα της δικαιοσύνης όπως ε, αυτή ασκείται στα διάφορα κράτη. Αυτό είναι ένα άλλος τρόπος, ένας άλλος τρόπος ώστε να είναι κανείς ε, Ευρωπαίος. Ορισμένοι επιμένουν για τη σημασία της εγγύησης στα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη να ανταποκρίνονται δηλαδή στα νομικά συστήματα αυτά όπως σας ανέφερα, που απόλυτα να είναι λειτουργικά. Την αρχή της δικαστικής συνεργασίας, την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία με τη σειρά τη βασίζεται στην μεγαλύτερη γνώση, βαθύτερη γνώση των διαφόρων συστημάτων. Και αυτό ακόμα είναι ένα στοιχείο το οποίο ήθελα να σας θυμίσω πως έχει ληφθεί υπόψη από τις τροπολογίες. Κάτι ακόμα, μια άλλη σειρά τροπολογιών που αφορούν τα διαδικαστικά δικαιώματα, δηλαδή την, στις ποινικέ διαδικασίες κυρίως. Οπότε ε, προτείνεται δωρεάν νομική αρρωγή και για τους ευαίσθητους κατηγορούμενους ή θύματα όπως επίσης και για την, το ένταλμα σύλληψης υπάρχουν προβλήματα. Τουλάχιστον εμείς από την Νομική Επιτροπή επιμένουμε γιατί ε, θα πρέπει στην Ευρώπη να λαμβάνεται παρκώς υπόψη η διαδικαστική, η διαδικαστική ε, πλευρά των δικαιωμάτων. Εμείς έχουμε συνηθίσει να ορίζουμε τα δικαιώματα του ουσιαστικά και αυτά περισσότερο γίνονται λάβαρα και όχι στη γεγονότα. Αλλά η διαδικασία είναι η εγγύηση για την εφαρμογή. Και έπειτα υπάρχουν διάφορες οριζόντες ενδιαφέροντες τροπολογίες που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κατά τη γνώμη μου ε, ήταν θετική αυτή η διοργάνωση κοινή συνεδρίασης για το πρόγραμμα της Οκάλμης και γιατί αυτό, γιατί σήμερα είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον όσο και η παραγωγή κοινών κανόνων στην Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό το να αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητά τους, η αποδοτικότητά τους. Δηλαδή να υλοποιούνται στην πράξη, να τίθεται σε εφαρμογή οι νομικές αρχές, οι ποινές, οι κυρώσει που ορίζονται από τον νόμο και να δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις όπως υπογραμμίζουν κάποιες τροπολογίες, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια πιο στενή συνεργασία ανάμεσα στην Κομισιόν, τα κρατημέλη και τις υπηρεσίες της διάφορης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή να μπορέσουμε έτσι περισσότερο να διαδώσουμε τις πληροφορίες σε σχέση με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών νομοθεσιών από πλευράς των κρατών μελών. Λοιπόν, ενημέρωση, όπως είπα, και εγγύηση της δυνατότητας παρακολούθησης, ανιχνευσιμότητας και άρα ε, εκ των ε, υστέρων αξιολόγηση και λειτουργικότητα του νομοθετικού συστήματος. Ορισμένες ε, τροπολογίες επίσης καλούν να δοθεί περισσότερη έμφαση στη δραστηριότητα παρακολούθησης της εφαρμογής, διότι το πρόβλημα της ελλειπούς εφαρμογής ή της του του, εξαιρετικού περιορισμού πραγματικών ε, στόχων ε, ε, είναι το πιο σημαντικό και προφανές πρόβλημα. Επ' αυτού παρεμβαίνει και ένα, μάλλον αναφέρεται και ένα άλλο σημαντικό έγγραφο που υποβλήθηκε στην Υπονομική Επιτροπή πριν από κάποιες μέρες και καλείται μελέτη από πλευράς του Policy Department μέσα για την εξασφάλιση της εφαρμογής και της αξιολόγησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, της αποδοτικότητας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ζητήσαμε λοιπόν μια τέτοια εργασία και ενισχύθηκε ε, η δική μας ε, βεβαιότητα για την σημασία και τη χρησιμότητα τέτοιων συνεδρίων μετά από τη δημοσίευση αυτού του εγγράφου από το Policy Department, το Τμήμα Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα σας αναφέρω κάποια πράγματα γιατί πρέπει να τα προσέξουμε όλα αυτά. Τίθεται ε, εντόνως το πρόβλημα ότι Παραδείγματο χάρη, όλε οι οδηγίε για το περιβάλλον δεν έχουν γίνει δεκτέ κατά 91%. Οι οδηγίες για την εσωτερική αγορά, για την ηθαγένεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα έχουν, έχουν γίνει δεκτές κατά 73%. Ε, μα τι κάνουμε εδώ πέρα και φτιάχνουμε κανόνες και οδηγίες άμα μετά δεν εφαρμόζονται ή δεν καν, ε, δεν μεταγράφονται. Καταλαβαίνετε τι τεράστια αντίφαση εδώ πέρα για με τη δουλειά που κάνουμε. Μας οδηγεί ως νομοθέτες στο ε, καθήκον, όχι μόνο να νομοθετούμε, αλλά να πετούμε από την Κομισιόν και από την ολόκληρη την Ένωση να κουνηθούν ώστε όλα αυτά που εμείς νομοθετούμε και κόντρα νομοθετούμε να πάρουν σάρκα και οστά και να περπατήσουν στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Παράδειγμα, έχει αυξηθεί ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάση και άρα υπάρχουν περισσότερες διαδικασίες απέναντι στα κράτη-μέλη που δεν είναι εντάξει. Και πρέπει να υπογραμμίσουμε πως ήταν θετικός αντίκτυπος του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ένωσης, διότι η μεταγραφή των οδηγιών ξεκινά, αρχίζει τουλάχιστον όσον αφορά την ταχύτητα της μεταγραφής. Όχι μόνο τη μεταγραφή, αλλά και την ταχύτητα της μεταγραφής η οποία αυξήθηκε από το 10% στο 24% στην τελευταία περίοδο που μελετάτε. Θα πρέπει λοιπόν να κατηργηθούν οι φραγμοί και τα εμπόδια για την ταχεία μεταγραφή των νομοθεσιών. Και αυτό προκύπτει και αυτό οφείλεται στην αοριστία με την οποία ε, η οποία μάλλον διέπει τις οδηγίες και το γεγονός ότι οι διοικητικές και νομικές διαδικασίες πολύ συχνά είναι περίπλοκες και πολύ αργές στο εσωτερικό των χωρών και οι διαφορές ερμηνείας αυξάνονται. Πολύ ανησυχητικά. Επιτρέψατε μου λοιπόν να επιμείνω ότι υπάρχει πρόβλημα εφαρμογής και πάνω απ' όλα μεταγραφής των οδηγιών. Και μετά μετατρέπεται και σε πρόβλημα επιβολής του νόμου. Και εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας. Αυτή η έκθεση η οποία παρουσιάζει το Policy Department, αυτή η μελέτη είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε την υπηρεσία από τη συνέταξη. Ωστόσο υπάρχει μια απόχρωση δίκαιη για τα στοιχεία παράβασης από πλευρά των κρατών μελών ή της αργής αποδοχής μεταγραφής. Όμως αυτό δεν αρκεί. Σήμερα πρέπει να προβληματιστούμε για κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα ξεκινήσει ή όχι επαρκώς ίσως από κάποιους ε, μελετητές, αλλά όχι από τα ίδια τα θεσμικά όργανα. Και τι σημαίνει αυτή, αυτός ο προβληματισμός, ότι πρέπει να καταλάβουμε αν η δυσκολία μεταγραφής εφαρμογής και άρα απόδειξης της, της ε, του νομοθετικού μας ε, πλαισίου οφείλεται στην αργή αποδοχή μεταγραφή από τα κράτη-μέλη ή οφείλεται και άρα μάλλον αν η θεραπεία είναι μόνο τιμωρία των κρατών μελών που αργούν ή, αν, ή μήπως το πρόβλημα είναι τελικά η ίδια η δομή των κανόνων που εγκρίνουμε, αλλά κυρίως η γνώση από πλευράς των πολιτών των δικαιωμάτων τους, η, δημιουργία μιας κοινή νομικής συνείδησης στην Ευρώπη. Ίσως αυτός να είναι ο άλλος λόγος. Και από αυτό νομίζω πως δεν έχουμε προετοιμαστεί επαρκώς, αλλά θα πρέπει νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση να προχωρήσουμε και γι' αυτό και θεωρώ και θυμίζω μια θετική πρωτοβουλία της Κομισιόν, δηλαδή την ε, εκπόνηση πινάκων επιδόσεων στο πλαίσιο της δικαιοσύνης, που θα πρέπει να επεκταθεί βεβαίως σε όλους τους τομείς της δικαιοσύνης και αυτή είναι μια πτυχή που υπογραμμίζεται από τις τροπολογίες. Και μια δική μου τροπολογία υπογραμμίζει πως τα νομικά συστήματα υψηλής ποιότητας μπορούν να παίξουν θεμελιώδη ρόλο στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ευρώπη και ότι οι αποφάσεις είναι δομικά στοιχεία της ε, εμπιστοσύνης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ε, ε, ηθαγένειας. Κλείνω με το νομικό, την νομική κατάρτιση. Κατάρτιση όλων των φορέων δικαίου. Η υλοποίηση του χώρου ελευθερίας και ασφάλειας απαιτεί από όλους τους, αφορά μάλλον όλους τους ε, επαγγελματίες του δικαίου και κυρίως τους δικηγόρους, διότι η σχέση ανάμεσα στον πολίτη και τον δικαιοσύνη ορίζεται από τον δικαστή, αλλά ξεκινά, αρχίζει να κινείται από το άτομο εμπιστοσύνης των πολιτών, δηλαδή τους δικηγόρους. Και σε αυτό το πεδίο είμαστε πίσω όσον αφορά την κατάρτιση αυτού του μεγάλου κομματιού. Η τεχνολογία δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί επαρκώς. Η προσβασιμότητα στις πηγές ε, τις ενημερωτικές για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο δεν αρκεί. Θα πρέπει λοιπόν να στηριχθεί η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αλλά και οι γλωσσικές πτυχές που πολύ συχνά έχουν υπογραμμιστεί από διάφορες τροπολογίες. Και αν προχωρήσουμε σε αυτές τις διορθώσεις, δεδομένου ότι έχουμε κάνει μια συνεδρίαση, μάλλον μια ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματος της Οκχόλμης σε σχέση με την αποτελεσματικότητά του θα πρέπει να δώσει αποτελέσματα τέτοιας φύσεως. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε κύριε Μπερλιγκουέρ και τώρα θα ακούσουμε τον Πρόεδρο της Επιτροπής ΑΦΚΟ, τον κύριο Κάρλο Καζίνη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, εγώ θα είμαι σύντομος. Θα ξεκινήσω από δύο οπτικές γωνίες που περιορίζουν τη σκέψη μου. Η πρώτη είναι ε, αυτή ε, που έδωσε περισσότερο η Επιτροπή ΑΦΚΟ, που είναι η Συνταγματική Επιτροπή. Θα μιλήσω δε για αυτούς τους, ε, αυτές τις οπτικές γωνίες. Πρώτον, της Συνταγματικής Επιτροπής και δεύτερον θα κάνω ένα γενικό σχόλιο για τις τροπολογίες που αφορούν, που μάλλον που έχουν υποβληθεί και που αφορούν, είναι πολυάριθμες, αλλά που δεν θα σας τις αναφέρω μία προς μία αλλά συνοπτικά. Ορισμένε τροπολογίε είναι τυπικέ, δηλαδή, φορούν δηλαδή τη διατύπωση και τι βρίσκουμε καλέ εφόσον βελτιώνουν το νόημα. Αλλά υπάρχουν άλλε τροπολογίε που αφορούν την ουσία, την, διεξουσία ε, του Κοινοβουλίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη θέση των Εθνικών Κοινοβουλίων, του εκλογικού νόμου Είναι θέματα τα οποία αφορούν άμεσα την Επιτροπή ΑΦΚΟ, η οποία επί όλων αυτών των θεμάτων έχει ήδη συζητήσει, έχει παρουσιάσει ψηφίσματα τα μεγάλο κομμάτι των οποίων, εκ των οποίων έχει ήδη υπερψηφιστεί. Όσον αφορά της εξουσίας του Κοινοβουλίου, είναι σαφές ότι εγώ πρέπει να εκφράσω αντίθετη γνώμη για όλες τις τροπολογίες που στόχο έχουν να περιορίσουν ε, τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Βασικά, πρόκειται για τροπολογίες που θέλουν να καταργήσουν τα όσα λέει η έκθεσή μας. Και είμαι κατά. Είμαι αντίθετα υπέρ όλων των τροπολογιών που με κάποιο τρόπο προσπαθούν να δείξουν ε, γραμμές βελτίωσης για τις δημοκρατικές εξουσίες και τις νομοθετικές εξουσίες του Κοινοβουλίου. Πρέπει δηλαδή να συνεχιστεί ο προβληματισμός για τη διαφάνεια που είναι απαραίτητη, ακόμα και όταν ε, γίνονται τριμερείς ε, διάλογοι που σήμερα σε μεγάλο βαθμό καταλήγουν και ξεπερνούν το γράμμα της συναπόφασης μέσω της πρώτης, δεύτερης, τρίτης ενδεχομένως επαφής. Ε, χρειάζεται ωστόσο περισσότερη διαφάνεια. Πιστεύω πως είναι σωστό να υπογραμμίσουμε την ανάγκη για μια πρωτοβουλία της Επιτροπής που να δέχεται πιο συχνά τα αιτήματα του ε, Κοινοβουλίου και με ενδεχόμενη αναθεώρηση των συνθηκών μια, ένα δικαίωμα πρωτοβουλίας είτε άμεσο είτε που δίνεται από το Κοινοβούλιο. Ε, υπάρχουν επίσης τροπολογίες που πρέπει να προσεχθούν ε, σύμφωνα με τις οποίες ε, θα πρέπει να πάψει η πρακτική των πολιετών προγραμμάτων όπου υπάρχουν επαρκείς νομικές βάσεις για να μπορούμε να εκδίδουμε ε, νομοθεσίες, να συντάσσουμε νομοθεσίες όπου συμμετέχει και το Κοινοβούλιο. Τώρα αφορά τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Σύμφωνοι είμαστε με τις περισσότερες τροπολογίες. ω Επιτροπή ΑΦΚΟ ασχοληθήκαμε περισσότερο με την προσχώρηση στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτή η συζήτηση. Υπάρχουν όμως προβλήματα που έχουν λυθεί και άλλα που δεν έχουν λυθεί. Και οι τροπολογίες μας παροτρύνουν να κλείσουμε αυτή την εργασία και να είμαστε και είμαστε έτοιμοι να τις δεχτούμε. Θα ήθελα να κάνω μόνο μια σύντομη παρατηρήση. Εγώ θα απέφευγα τις απαριθμίσεις ε, των διαφόρων περιπτώσεων διάκρισης. Κάθε περίπτωση διάκρισης κατά ενό ανθρώπου έναντι άλλου ανθρώπου είναι σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι νομικοί τα γνωρίζουν όλα αυτά. Ε, ε, κατά τη γνώμη μου λοιπόν αρκεί μια σαφής σταθερή υπόδειξη πως είναι κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας οποιαδήποτε διάκριση για οποιαδήποτε κατηγορία ανθρώπου. Τώρα, Όσον αφορά το θέμα των Εθνικών Κοινοβουλίων, υπάρχουν τροπολογίες που θέλουν να εισάχουν ένα είδος ελέγχου της επικουρικότητας για την περιφερειακή νομοθεσία, όχι μόνο την κρατική νομοθεσία. Δηλαδή, έλεγχο όχι μόνο κρατικό αλλά και περιφερειακό για το, ε, στο όνομα της επικουρικότητας επί των επί της νομοθετικής δραστηριότητας του Κοινοβουλίου. Νομίζω πως αυτό σημαίνει αλλαγή των συνθηκών και άρα δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. Ωστόσο προσωπικά θα μπορούσα να το συζητήσω, αλλά είμαι κατά. Πολλές ε, τροπολογίες δεν αναφέρονται στον εκλογικό νόμο. Και εδώ δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτό που μας ε, ζητούσε η συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν φτιάξαμε δικό μας εκλογικό νόμο. Περιοριστήκαμε σε κάποιες προσαρμογές γραφειοκρατικού χαρακτήρα, αλλά δεν κάναμε πολλά από αυτά που μας ζητήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει είμαι κατά της νομοθεσίας από τη στιγμή που δεν μιλάνε για ομοιόμορφο εκλογικό νόμο γιατί είναι αυτό κατά της συνθήκης και άρα οδηγεί σε μια σκεπτικιστική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αντίθετα, θα πρέπει να επιμείνουμε για την ιδέα μιας ομοιόμορφης, ενός ομοιόμορφου εκλογικού νόμου προς όφελος της διαφάνειας για την επιλογή των υποψηφίων από πλευρά των κομμάτων, αναζήτηση ενό κριτηρίου, μια μαθηματική φόρμουλα, σε πάση περιπτώσει, ε, που να μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να μπλεχτούμε σε ένα συζητήσεις για το ποιος μπορεί και πόσοι θα είναι μάλλον οι βουλευτές για κάθε φορά που θα μπαίνει άλλη μια χώρα, όπως έγινε με την Κροατία. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα συγκεκριμένος αριθμός και τέρμα και η συζήτηση γι' αυτό. Τώρα, για τις περιφερειακές ε, εκλογές, ε, κάποιες τροπολογίες ζητούν την άμεση εκλογή σε ευρωπαϊκά αξιώματα. Ήδη εκφράσαμε θετική άποψη όσον αφορά το πρόεδρο της Επιτροπής. Γι' αυτό δεν υπάρχει θέμα. Πρέπει όμως να σκεφτούμε και να συζητήσουμε άλλα ζητήματα που αφορούν τους ε, μεμονωμένους επιτρόπους ή άλλα αξιώματα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν έχουμε επίση τίποτα να πούμε, παρά μόνο να είμαστε θετικοί απέναντι σε αυτό που κατά κάποιο τρόπο πρότεινε η ΑΦΚΟ όσον αφορά την υπέρβαση των γραφειοκρατικών εμποδίων στη συμμετοχή, τη δραστήρια στην Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκές εκλογές, ιδιαίτερα όσον αφορά τους πολίτες, τους Ευρωπαίους που κατοικούν σε διαφορετικές χώρες από τις χώρες προέλευσής τους, η εθνικότητάς τους. το οι άλλε τροπολογίε ε, σχετίζονται με την πρωτοβουλία των πολιτών που θα έπρεπε να είναι μία από τι ε, μεγάλε καινοτομίε, τι κύριε καινοτομίε τη ε, συνθήκη τη Λισαβόνα. Ω προ αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, αλλά χρειάζεται να προσεχθεί περισσότερο. Δηλαδή δεν μπορούν να, γίνουν δεκτέ όλε οι πρωτοβουλίε. Υπάρχει και οικονομικό θέμα οι πολίτε για να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη μορφή άμεσης δημοκρατίας χρειάζεται να ε, στηρίζονται οικονομικά με κάποιο τρόπο διαφανή. Δυστυχώς όμως και υπογραμμίζεται εδώ δικαίως σε κάποιες τροπολογίες πως η τάση του συστήματος ε, για συλλογή ηλεκτρονικών πληροφοριών είναι εξαιρετικά περίπλοκη και δαπανηρή και άρα χρειάζεται να παρέμβουμε για να καταστεί πιο εύκολη η πρόσβαση. Πρέπει ωστόσο να προσέξουμε να μην γίνεται για ψήλου πίδημα αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών, εάν δεν υπάρχει δηλαδή κανένας έλεγχος. Αυτό σημαίνει κάποιες ε, ε, κάποια περίπλοκο χαρακτήρα δεν μπορεί να απλοποιηθεί παντελώς, ωστόσο να καταστεί πιο εύκολη η συμμετοχή. Και ίσως θα ήταν δίκαιο να, να σκεφτούμε στην επόμενη θητεία τις επιπτώσεις των πρωτοβουλειών που ανταποκρίνονται στο στόχο μας. Τον αριθμό δηλαδή των υπογραφών. Αν και θα πρέπει να αριθμίζονται καλύτερα αυτές οι πρωτοβουλίες. Στην πράξη, και τα είπα όλα όσα αφορούν τις εργασίες της Επιτροπής της οποίας προεδρεύω. Θα ήθελα μόνο να εκφράσω μια θετική γνώμη για κάποιες πτυχές που αντίθετα μας, βλέπουν, ε, ε, μας βρίσκουν μάλλον ε, μας καλούν μάλλον το ενδιαφέρον, αλλά δεν είμαστε αρμόδιοι. Όπως ας πούμε το θέμα της μετανάστευση και του ασύλου, που σε όλε τι τροπολογίε που υποβλήθηκαν στόχο έχουν να στηρίξουν εκείνους που προτείνουν μια ισορροπία ανάμεσα στην απέτηση ασφάλειας, τη σεβασμό της νομοθεσίας αλλά και τη φιλοξενία. Κυρίως επί τη βάση της αρχής για την οποία έχω επιμείνει επανειλημμένος, όχι μόνο γιατί με ενδιαφέρει ως Ιταλό, και άρα πολίτη ενό κράτου μέλου που μαζί με άλλα κράτη της Νότιας Ευρώπη ενδιαφέρονται ιδιαίτερα γιατί καθημερινά, καθημερινά ε, έχουν να αντιμετωπίσουν τη μετανάστευση αλλά και επειδή μου φαίνεται πω είναι μια αρχή λογική ε, συνεπή με την ευρωπαϊκή ιδέα ότι τα σύνορα της, Ελλάδα, τη Ιταλία, τη Ισπανία, τη Μάλτα Μάλτας ε, και τα λοιπά δεν είναι μόνο εθνικά σύνορα αλλά είναι κυρίω ευρωπαϊκά όνειρα και εφόσον έχουμε ενωμένη Ευρώπη Ας το αναλάβει η Ενωμένη Ευρώπη αυτό το πρόβλημα. Με μορφές παρέμβασης που να είναι συνεπείς και συνεκτικές και για την ασφάλεια και για την υποδοχή των ε, μεταναστών. Συμφωνώ επίσης ε, για τα θέματα που προτείνονται στα θέματα δικαιοσύνης και ιδιαίτερα τα όσα είπε ο συνάδελφος Μπερλιγκουέρ για την ανάγκη της ε, κατάρτισης των εισαγγελέων και δικηγόρων και νομικών γενικότερα και όσον αφορά τα δικαιώματα τα διαδικαστικά. Ε, <clears throat> αυτά τα είπε ο Μπερλιγκουέρ, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πρόεδρε Κασίνη και τώρα αν μου επιτρέπετε ως εισηγητής εξ ονόματος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρουσίαση της δικής μου θέσης σε σχέση με τις ε, τροπολογίες που έχουν παρουσιαστεί σε σχέση με τα θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Εν συντομία, θα ήθελα να αντιμετωπίσω τα εγκάρσια θέματα. Δηλαδή, τα θέματα που έχουν οριζόντιο χαρακτήρα και τα οποία αναφέρονται σε πάρα πολλές τροπολογίες. Είναι πολλές βέβαια οι τροπολογίες, πάνω από 300. <clears throat> Πρώτα απ' όλα θέλω την υποστήριξή σας ώστε η έκθεση αυτή που θέλουμε να συντάξουμε να είναι συνοπτική και σύντομη, να έχει σαφή μηνύματα και να εστιάζεται στην εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης. Για το λόγο αυτό δεν θεωρώ ότι ευσταθούν οι τροπολογίες οι οποίες ε, συζητούν και θέλουν να τροποποιήσουν ορισμένα πράγματα για τα οποία ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια σταθμισμένη και δημόσια άποψη όπως η είσοδος στην περιοχή του Σέγγεν της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Πολλές από αυτές τις τροπολογίες λοιπόν ταυτίζονται και θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εκπόνηση τροπολογιών συμβιβασμού για αυτές τις τροπολογίες, κάποιες από τις οποίες όπως είπα είναι πιο σχετικές με το θέμα από ότι ορισμένε άλλες το θέμα της εξωτερικής διάστασης του χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας είναι κάτι που είναι σημαντικό. Πιστεύω και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Άλλες τροπολογίες αναφέρονται σε ιδιαίτερα θέματα και όταν περάσουμε στην σύνταξη τροπολογιών συνασπισμού, εγώ θέλω να διατηρήσουμε την εστίαση στις λεγόμενες πόλεις ιέρειας, στις περιοχές που έχουν να κάνουν με τη χάραξη πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλε τροπολογίε αναφέρονται στην εκλογική νομοθεσία. Εδώ δεν νομίζω ότι είναι η, η δική μας ε, απόλυτη αρμοδιότητα, αλλά θα συζητήσω με τους συναδέλφους ώστε να υπάρχει και κάποια μνήμα των θεμάτων αυτών στην τελική σύνταξη. Επίσης, <clears throat> πιστεύω ότι το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει να δρουν λαμβάνοντας υπόψη το νέο θεσμικό στερέωμα που δημιουργήθηκε με τη Σύνθηκη της Λισαβόνας όπως γνωρίζουμε όλοι μας έχει μια ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του Κοινοβουλίου στην ανάπτυξη του χώρου ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας και γι' αυτό η ειδική μου τροπολογία 4 είχε σαν στόχο να αναφερθεί συγκεκριμένα και εκπεφρασμένα στην σημασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την προστασία τους και στην συμπληρωματικότητα αυτής της προστασίας με τα εθνικά νομικά πλαίσια. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δώσει σε όλους τους πολίτες το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας, όπως λέει το άρθρο 53 της Ευρωπαϊκής Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που είναι προσαρτημένη στην Συνθήκη της Λισαβόνας. Πολλοί συνάδελφοι έχουν καταθέσει τροπολογίες που αναφέρουν ότι θα πρέπει να αναφέρεται το πρόγραμμα της Λισαβόνα σε μια πιο περιεκτική ευρωπαϊκή ηθαγένεια, όχι μόνο δηλαδή τους πολίτες των κρατών μελών, αλλά και αυτούς που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους μετανάστες. Ότι λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να αφορούν όλους αυτούς που βρίσκονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το καθεστώς ηθαγένειάς τους. Επίσης, αυτό το οποίο ήταν στο παρελθόν διακυβερνητικού χαρακτήρα τα προγράμματα της Χάγης και του Τάμπερε και αυτό ίσχυε και με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Όλα αυτά έχουν περάσει με την ε, εφαρμογή τη συνθήκη τη Λισαβόνα σε ένα ενωσιακό πλαίσιο. Έχει η Κομισιόν λοιπόν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα τη πρωτοβουλία σε τομεί που τώρα καλύπτονται από αυτό για να προωθήσει περαιτέρω το πρόγραμμα της Στοκχόλμης μια σημαντική διάσταση του νέου αυτού χώρου ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας είναι και η σύνδεση με τα εθνικά κοινοβούλια, κάτι το οποίο το υποστηρίξαμε σε όλη τη διάρκεια της θητείας μας. Θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη συνάρθρωση με την πρακτική με τα εθνικά κοινοβούλια στα πλαίσια της ε, επικορικότητος και με πλήρη σεβασμό του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων. οι εκπρόσωποι των πολιτών και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο έχουν, μια, έχουν αντίστοιχες προκλήσεις να αντιμετωπίσουν. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να έχουμε ένα συνεκτικό πλέγμα ε, δραστηριοτήτων όπου θα συμμετέχει και το Συμβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφέρεται επίσης το λεγόμενο δίλημα της Κοπεχάγης στις ε, τροπολογίες. Κάτι που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές σε, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Είναι απαραίτητο ο πίνακας επίδοσης για τη δικαιοσύνη να δίνει σημασία και στο επίπεδο ποιότητα στο οποίο εφαρμόζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ίδιο σε σχέση με την αναζωπήρωση του λαϊκισμού, του εξτρεμισμού, της ξενοφοβίας κτλ. που αναφέρονται σε πολλές τροπολογίες από την Επιτροπή Λίβε. Είναι σαφές ότι το νέο αυτό πρόγραμμα θα πρέπει να λάβει υπόψη του ιδιαίτερα τα προβλήματα αυτά, να αντιμετωπίσει την ξενοφοβία, τον στιγματισμό των ε, διαφορών, τις προκαταλήψεις εναντίον ορισμένων ε, πολιτών μας, την ε, μυσαλλοδοξία, όπως έγινε σαφές από την πρόσφατη ακρόαση της Επιτροπής Λίμπερ. Επίσης ε, η τροπολογία μου 102 αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων να αποχωρήσει λοιπόν το η μέτρων για τα προσωπικά δεδομένα. Βρισκόμαστε προς το τέλος της θητείας μας, επομένως δεν μπορούμε να αφήσουμε να χαθεί αυτή τη τόσο σημαντική πτυχή για τους πολίτες μας. Θα ήταν ένα πολύ σοβαρό σφάλμα σε ό,τι αφορά τον απολογισμό τις δράσεις του Κοινοβουλίου μας και υπήρχαν επίσης και κάποιες τροπολογίες σε ό,τι αφορά τα δικονομικά δικαιώματα και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο όπου υπάρχουν ακόμα κάποια τεχνικά στοιχεία τα οποία πρέπει να συζητηθούν περισσότερο το ίδιο σε ό,τι αφορά τη στρατηγική εσωτερική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταία ολομέλεια εγώ έκανα μια προφορική ερώτηση στην Κομισιόν που οδήγησε σε συζήτηση και σε ψήφισμα. Το περιεχόμενο αυτού του ψηφίσματος λοιπόν θα πρέπει να αντανακλάται και αυτό στην τελική διατύπωση της έκθεσής μας σε σχέση με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Επίσης έχω την τροπολογία 254 που ζητά ότι η διαχείριση των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτό να γίνεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και από τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι <clears throat> θα πρέπει και στην εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνεται υπόψη και η διάσταση του κράτους δικαίου, των πολιτικών ασύλου και το να υπάρχουν κοινέ πολιτικές ασύλου και παροχής καταφυγίου στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά σύμφωνα με αυτά που άκουσα από τον Κάλο Κασίνη και τον Λουίτσι Μπελίνγκουερ σε σχέση με τη δυνατότητα, με τη σημασία που έχει μια νομική κουλτούρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τονίσει πάντα στις συζητήσεις αυτές ότι δεν μπορεί να είναι μονάχα θεσμικού χαρακτήρα η εφαρμογή του προγράμματος Στοχόλμης. Δεν πρέπει να καταλαμβάνει μονάχα τους θεσμικούς παίκτες, αλλά πρέπει όλοι οι νομομαθείς και οι δικηγόροι και οι δικαστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συμμετέχουν πλήρως για να μπορέσει να επιτευχθεί το σύνολο αυτών των ε, ε, φιλοδοξιών του προγράμματος της Χολμς με το να είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο δικαστικό τομέα καλύτερα ε, γνώστες της ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών πολιτικών. Όλα αυτά λοιπόν δεν πέφτουν από τα δέντρα όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες, όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με υποστήριξη προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε όλοι οι επαγγελματίες του δικαίου στην Ευρώπη να ξέρουν ακριβώς ότι είναι απαραίτητη και δική τους ε, βοήθεια και ε, συμβολή στην εφαρμογή της δικαιοσύνης. Όλοι μας λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε αυτή την ευκαιρία μιας καλύτερης συμμετοχής έναντι της... Ε, ε, ε, κύριε, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ενδεχομένως θα ήθελε να λάβει λόγο τώρα και να παρουσιάσει την απόψή του και η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι παρούσα, αλλά επίσης έχουμε και μια σειρά από κοινοβουλευτικούς οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο και δίνω καταρχήν το λόγο στον κύριο Γκερέρο Σαλόμ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω φυσικά να ευχαριστήσω τους τρεις εισηγητές για τη δουλειά τους. Γνωρίζουμε όλοι πόσο πολύπλοκο είναι να εργάζεσαι με όχι ακριβώς την ίδια προοπτική ε, και πρόκειται για την ίδια έκθεση, κοινή έκθεση. Εγώ κατέθεσα αρκετές τροπολογίες. Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων μεταξύ των τριών είναι αυτή η οποία έχει καταθέσει τις λιγότερες τροπολογίες. Ε, έχει μια λογική και αυτό. Ο κύριος Κασίνη πρόεδρος Επιτροπής μας ε, έκανε μία αναδρομή σε αυτές τις τροπολογίες περισσότερες εξ αυτών. Γι' αυτό και εγώ θα είμαι πάρα πολύ περιεκτικός, περιληπτικός. Και θα πω ότι ναι, μεν προέρχονται από την Επιτροπή ΑΦΚΟ και από ένα μέλος Επιτροπής ΑΦΚΟ, αλλά δεν έχουν ε, θεσμική εστίαση θα έλεγα, αλλά ε, στο επίκεντρό τους βρίσκονται οι πολίτες. Όταν καταθέτουμε παραδείγματος χάρη για την πρόσβαση στα έγγραφα, ενισχύουμε όχι μόνο τη διαφάνεια, που θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μια θεσμική συμπεριφορά, αλλά και το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσα στον οποίο λαμβάνονται και οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητάμε να ενισχυθεί ο ρόλος της Κομισιόν να έχει ηγετική θέση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι που βλέπετε από τι συνθήκε. Άρα, ουσιαστικά τι ζητάμε με αυτό, προστασία των πολιτών μέσω αυτή τη παρέμβαση τη Κομισιόν ή όταν λέμε ότι είναι ανάγκη να γίνει μνήμα. Ε, στο καθεστώς ε, των κομμάτων, καταστατικών κομμάτων και ιδρυμάτων, ουσιαστικά προασπιζόμαστε το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πολιτική συμμετοχή, συμμετοχή στα πολιτικά δρόμενα μέσω των κομμάτων ή μέσω των ε, ιδρυμάτων. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι γίνεται πολλής λόγος στο εκλογικό σύστημα. Το είπε και ο κύριος Κασίνη και ο κύριος Λόπεθα Γιλάρου. Είχαμε μία μακρά αλλά αποτυχημένη, καθόλου καρποφόρα διαδικασία, όχι στο πλαίσιο της ΑΦΚΑ, αλλά συνολικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κακό να ζητήσουμε τουλάχιστον αυτό κάνω εγώ με μια τροπολογία μου, να προχωρήσουμε σε ένα δικό μας αυτόνομο εκλογικό σύστημα που θα είναι όλο και πιο ομοιογενές, όλο και πιο ομοιόμορφο. Ο όρος βέβαια ομοιόμορφο ή ομοιογενές είναι ένας όρος που δημιουργεί πρόβλημα και δεν το αναφέρουμε, αλλά αν αναφέρθουμε σε ένα ίδιο σύστημα που θα ρυθμίζει σε που θα είναι αυτόνομο δηλαδή αυτό το σύστημα, από καθαρμένο από τα κλικά συστήματα των εθνικών κρατών που μπλοκάρουν τις τροποποιήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλο και πιο ομοιογενές, να μην είναι δηλαδή ακριβώς το ίδιο παντού, αλλά να έχει κοινά στοιχεία ώστε οι πολίτες να μπορούν να έχουν την πολιτική συνείδηση ότι όταν ψηφίζουν σε ευρωεκλογέ ψηφίζουν ε, κάτι ε, συγκεκριμένο και όχι, δεν, δεν πρόκειται για μια προέκταση των βουλευτικών ή των δημοτικών εκλογών. Ευχαριστώ πολύ κύριο Λούχαν, λέει ο Πρόεδρος. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα αγαπητοί συνάδελφοι, Θέλω να ευχαριστήσω τους τρεις εισηγητές για την πολύπλοκη αλλά πλήρη αυτή έκθεση που πραγματεύεται θέματα πολλά και ευαίσθητα, λεπτά θέματα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. ιδίω ό,τι αφορά τι χώρε που είναι ακόμα σε μεταβατική φάση, δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει ή μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο όλη αυτή την νομοθεσία. Υπάρχουν ε, βέβαια ακρός πολύπλοκα ζητήματα ε, που δεν μπορούμε να τα καλύψουμε τώρα ε, αναλυτικά. Αλλά θα πρέπει στην Επιτροπή ΛΥΠΕ και στο Κοινοβούλιο εν γέννη ή και τα άλλα θεσμικά όργανα να ε, αναφερθούμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, την ηλεκτρονική ψηφοφορία συγκεκριμένα, που είναι ένα δικαίωμα για τον Ευρωπαϊκό πολίτη και εδώ διαπιστώνουμε ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα. Διότι σε ορισμένα μέλη, οι πολίτε δεν μπορούν να, να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Κατά την άποψή μου, είναι μια πτυχή αυτή που θα πρέπει να ρυθμιστεί και μάλιστα άμεσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι ρόλο έχει όταν λέμε ότι τις εκλογές δεν ρυθμίζουν τα μελη Θα έπρεπε να κάνουμε ε, μια συζήτηση πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, να διατυπώσουμε προτάσεις. Ένα δεύτερο θέμα για το οποίο θα σας μιλήσω είναι η διαδικαιοσύνη. Ο ορισμός Τη δικαιοσύνη από μια χώρα στην άλλη διαφέρει. Όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, για την υπεράσπιση ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μιλάμε για τη δικαιοσύνη ουσιαστικά. Η δικαιοσύνη... Είναι ένα φύλακα, ένα φρουρός που βλέπει τι πάει και τι δεν πάει καλά. Και στο οικονομικό επίπεδο μεταξύ άλλων. και στον τομέα της υπανόρθωσης οικονομικών αδικημάτων ή αδικιών και εκεί είναι ε, λιματική δικαιοσύνη θα έλεγα. Έχουμε ποινές θερητικές ελευθερίας σε κάποια συστήματα ε, για τα άτομα τα οποία έχουν διαπράξει αξιόπινες, πράξεις. Όμως σε πολλά συστήματα, σε πολλά ε, συστήματα δικαστικό όπως και στη δική μου χώρα, δεν δίνεται παρκής προσοχή στο ζήτημα της ε, επανόρθωσης ε, οικονομικών απολειών για αποκατάσταση οικονομικών ε, ζημιών απολειών. Δεν προβλέπεται παραδείγματος χάρη πρόστιμο για ανάκτηση των ποσών για τα που δεν φορολογήθηκαν σε περιπτώσεις δηλαδή φοροαποφυγής ή φοροδιαφυγής. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε αυτά τα θέματα να τα συζητήσουμε. Για να δούμε μήπως θα μπορούσαμε αυτήν την έννοια της δικαιοσύνης να την αναδιοργανώσουμε, αν μπορώ να το πω έτσι. Να έχουν δηλαδή τα κράτη οικονομικά ωφέλη ή πλονεκτήματα στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή φόρο αποφυγής. Και ένα τελευταίο πολύ ενδιαφέρον για τη δική μου χώρα σημείο είναι και καταθέσαμε και πολλές τροπολογίες ε, σχετικά είναι ο χώρος Σέγγεν. Μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα, μιλάμε για κοινά δικαιώματα, για το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία, για την εσωτερική αγορά ή την κοινή αγορά. Ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε και για μία κατηγορία πολιτών ε, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία και μόνη, και να μην ε, δημιουργείται εντύπωση ότι κάποιοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας ή με περιορισμένα δικαιώματα για κάποιους λόγους. συμμετοχή στο χώρο Σέγγεν δεν ε, αποφέρει πολλά οικονομικά πλεονεκτήματα ή άλλου πλεονεκτήματα. Η συμμετοχή στο χώρο Σέγγεν είναι ένα ε, σημάδι εμπιστοσύνη και ισότιμη μεταχείριση όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Κάτι που χαρακτηρίζει το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, σεβαστείτε το χρόνο. Αλλιώ θα έχουμε προβλήματα με του διερμηνεί. Έχουμε χρόνο μόνο μέχρι τι 12.30. Ίσως μπορούμε να έχουμε κάποια λεπτά ακόμα. Κυρία Ρομέρο Λόπεχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα απλώ να αναφερθώ στη σημασία που έχει αυτή η ενδιάμεση έκθεση την οποία εκφωνούμε και ελπίζω ότι αυτές οι προτάσεις θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε μια τελική αξιολόγηση. Πρόκειται μονάχα για την πρώτη φάση του προγράμματος της Στοχόλμης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε πολλές επιτροπές μαζί. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχει το πάντα σαν βάση την ε, συνδίκηση Λισαβόνα και τα θεμελιώδη δικαιώματα και επίσης και η Συνταγματική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αγωνιστεί για αυτά τα θέματα. Θέλω να υπογραμμίσω λοιπόν αυτή τη, συμ... τη σημασία της ισορροπίας που θα πρέπει να υπάρξει σε ό,τι αφορά τη θεμετολογία αυτής της ενδιάμεσης έκθεσης και θα ήθελα να σας κάνω τώρα μία πρόταση. Μιλάμε για μία στατηγική εσωτερικής ασφάλειας για το 2014. Αλλά δεν μιλάμε για μία ε, στατηγική για την εδραίωση και την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό όσο η εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν τόσες πολλές ανισομέρειες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και σε επίπεδο προϋπολογισμού. Γιατί οι προϋπολογισμοί πάντα πηγαίνουν για να αντιμετωπίσουν τις απειλές ή τις υποτιθέμενες απειλές. Υπάρχουν λοιπόν πολλά να συζητηθούμε και χαίρομαι που γίνεται αυτή η συζήτηση σε επίπεδο ενδιάμεσης έκθεσης. Κυρία Λίχτενμπεργερ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα εγώ να σας τονίσω και πάλι πόσο σημαντική είναι η συμπερίληψη και του νέου ε, εργαλείου για την εποπτεία της εφαρμογής του ισχύοντος δικαίου στα κράτη-μέλη. Γιατί αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι οι κανόνες της ελεύθερης διακίνησης εφαρμόζονται με πολύ με διαφορετικό τρόπο στα κράτη-μέλη. Πολλές φορές καθυστερεί η εφαρμογή ή αλλοιώνεται ή εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο και αυτό δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα είναι η εξασφάλιση των δικονομικών δικαιωμάτων σε ποινικέ δίκες. Έχουμε τονίσει την ανάγκη να υπάρχει πρόσβαση σε μετάφραση και διερμηνία, προστασία των δικαιωμάτων, όλα αυτά. Όλα αυτά φυσικά θα πρέπει να οδηγήσουν σε καλύτερη στη συνεργασία των δικαστικών αρχών και καλύτερη κατάρτιση του δικαστικού προσωπικού. Αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν οι βάσεις για να υλοποιηθεί αυτό όπως έχουμε υποσχεθεί στους πολίτες ώστε να μπορεί κανείς να εγκαθίσταται όπου θέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν έχει δικαστικά προβλήματα <clears throat> θα έχει να αντιμετωπίσει ένα δικαστικό σύστημα το οποίο είναι προσιτό και προσβάσιμο στον πολίτη και μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλειά του ανεξάρτητα από τα εθνικά σύνορα. Κύριος Μπρόντς. Ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπερλενκουέρα για τα στοιχεία τα οποία μας αποκάλυψε ε, για το πόσο αργούν τα κράτη-μέλη να μεταγράψουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η Βρετανική μετάφραση μου είπε ότι είπατε πως πρέπει να ε, παταχθούν τα κράτη τα οποία ε, καθυστερούν και να δούμε και ποιοι είναι αυτοί που καθυστερούν. Μιλάτε όμως προσοχή γιατί μιλάτε λίγο για τα κράτη-μέλη σαν να είναι άτακτα παιδιά. Ε, και επίσης με πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε τον κύριο Κασίνη ότι θα πρέπει να απαγορεύεται κάθε διάκριση και όχι απλά ένας κατάλογος διακρίσεις επί τη βάση πολιτικής ε, γνώμης ή προς, η προσχώρηση, γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ενδυμική αυτή η κατάσταση και υποστηρίζεται από ολόκληρη την πολιτική τάξη. Ο κύριος Κασίνη μίλησε για την πρωτοβουλία μιας μορφής άμεσης δημοκρατίας. Υπάρχουν κάποιες επιφανειακές ε, ομοιότητες, αλλά βασικά είναι μόνο επιφανειακές, γιατί οι πρωτοβουλίε των πολιτών αντικατοπτρίζουν τη γνώμη αυτών που υπογράφουν και όχι την πλειοψηφία των ανθρώπων, των λαών και έπειτα δεν αποφασίζεται κάτι για το κράτος μέλος, είναι μια έκκληση για δράση από πλευρά της Κομισιόν που μπορεί κάλλιστα να το αρνηθεί. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν πιο πολλά κοινά ε, με τις αναφορές και όχι με τις αποφάσεις μιας άμεσης δημοκρατίας. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι αυτές οι αναφορές θα πρέπει να στηρίζονται οικονομικά. Επίσης γιατί υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε αυτές που θα εγκρίνονται και αυτές που θα, θα απορρίπτονται. Και επίση η Κομισιόν θα, είναι στην, ε, θα έχει να ε, διακρίνει κατά πόσο τα χρήματα αυτά προέρχονται από ε, ανεξάρτητους ή από τον ίδιο τον αναφερόμενο στις αναφορές. Έπειτα δεν έχουμε δυνατότητα Λέτε εδώ επίσης για το opt-out. Τι είναι opt-out και τι δεν είναι. Πρέπει να υπάρξει διευκρίνηση για όλα αυτά. Κύριε Βεσάριλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα ψηφίσαμε τη γνωμοδότηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, δική μου γνωμοδότηση, μουσκιώδης. Και θα ήθελα να πω ότι η γνωμοδότηση αυτή ε, εγκρίθηκε οι περισσότερες ε, δε τροπολογίες ε, είχαν ως στόχο τα δικαιώματα των μεταναστών για τα οποία έκανε ο κύριος Κασί να λαμβάνονται υπόψη ε, τα δικαιώματά τους. Αυτές ήταν οι περισσότερες τροπολογίες. Να σας πω βέβαια ότι δεν καταφέραμε να συντάξουμε πολλές συμβαστικές προτάσεις πλην μίας για τα θύματα τρομοκρατίας, επίσης και θύματα σωματεμπορίας, ε, για τους ανηλίκους. Έχουμε μια τροπολογία και ελπίζω να συνεχίσουμε και εσείς να συνεχίσετε να επεξεργάζεστε και να λάβετε υπόψη και τις σχέσεις τροπολογίες για τη στήριξη, προστασία, ε, την υποστήριξη των θυμάτων, εγκλημάτων κτλ. Μία πολύ σύντομη ερώτηση για το εκλογικό νόμο. Μιλήσατε για περιφερειακά και τοπικά και εθνικά συστήματα, κύριε Κασίνη. Γίνεται λόγο στην έκθεση όμως και για ευρωπαϊκό εκλογικό νόμο. Έρχονται ευρωεκλογέ. Θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε ε, για κάτι τέτοιο. Θα το αφήνατε έξω ή πιστεύετε πρέπει να το εξετάσουμε. Πριν στραφώ στους εισηγητές ξανά, από ό,τι βλέπω, ε, αντιλαμβάνω το Συμβούλιο δεν θέλει να σχολιάσει αυτή τη φάση. Μήπως θέλει Κομισιόν Σύντομα να πει κάτι. Πάρα πολύ σύντομα όμως παρακαλώ. Για να μην μας τελειώσουν οι διερμηνείς. Yes, thank you very much. Um, just very briefly and... Uh, ναι, πολύ σύντομα και σε αυτή τη φάση της συζήτησης η Κομισιόν Θέλει μόνο να, να επαναλάβει, επειδή υπήρξαν κάποιες τροπολογίε, προτινόμενε τροπολογίε, στην παράγραφο 5 του κειμένου ω έχει, θα θέλαμε να επαναλάβουμε τα όσα ήδη είπατε, κύριε Λόπες Αγγελά, ότι όλη αυτή η υπόθεση θα πρέπει να θεωρηθεί ε, ε μέσα στο πλαίσιο του νέου, του νέου θεσμικού πλαισίου θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια ε, όρημη και κανονική φυσιολογική πολιτική της Ένωσης. Η Κομισιόν να αποφύγει τους διάφορους καταλόγους στο μέλλον και να μην περιορίσει τις αρμοδιότητες του περχόμενου Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Άλλος από την Κομισιόν θέλει να μιλήσει. Παρακαλώ σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω απλά να τονίσω το ότι η έκθεση ζητά από την Κομισιόν να φτιάξει μια ευρωπαϊκή ε, ε, ένα σώμα αφύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων. Εδώ δεν μπορούμε να δεσμευτούμε, όπως δεσμευτήκαμε με το Frontex και το σχετικό κανονισμό που θα είναι στη διάθεσή σας μέσα στον επόμενο χρόνο. Να ε, αναφέρω λεπτομερείς στατιστικές για την καταπολέμηση του εμπορίου, του, του, του λαθρεμπορίου. Ε, ήδη κάνουμε πολλά. Είμαστε σε πολύ καλή βάση για τη συλλογή των στοιχείων, καθώς και για τη συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες. Η Κομισιόν τέλος θα υποβάλει ανακοίνωση για τις νέες προκλήσεις στο ε, δικαιοσύνη και στις εσωτερικές υποθέσεις και εδώ προγραμματιζόμαστε για το θέμα της αξιολόγησης και συμμεριζόμαστε τα όσα είπε ο κ. Μπελιγκουέρ για τη σημασία της αξιολόγησης, ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον. Ευχαριστώ και οι τρεις εισηγητές έχουμε σημειώσει όλα τα σχόλια που έγιναν. Ίσως ε, έγινε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση στον κύριο Καζίνη όσον αφορά το εκλογικό σύστημα, τον εκλογικό νόμο. Θέλετε να σχολιάσετε εν συντομία για να κλείσουμε παρακαλώ. Ναι, να πω σύντομα ότι συμφωνώ με τον συνάδελφο Γκουερέρο που είπε πως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια ομοιόμορφη, ένα εκλογική νομοθεσία σε αυτή την ψηφοφορία, θα αφήσουμε για την επόμενη. Συμφωνώ όμως με τον Γουερέρο ότι πρέπει να δοθούν κάποιες υποδείξεις για έναν εκλογικό νόμο, ότι θα πρέπει να υπάρξει, να είναι ομοιόμορφος, να είναι ισόρροπος και να αφορά όλα τα κράτη. Έχουν γίνει κάποια πράγματα, πρέπει να γίνουν κι άλλα. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και για τη συντομία σας. Ο κύριος Μπέλεγκουγκουέρ δεν έχει να προσθέσει κάτι. Οπότε κλείνουμε. Να ανακοινώσω μόνο, μόνο να ανακοινώσω ότι η... η μέρα που προβλεπόταν για την ψηφοφορία 21 Οκτωβρίου δεν γίνεται να γίνει ψηφοφορία τότε. Οπότε αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βρούμε άλλη ημερομηνία για την ψηφοφορία επί των τροπολογιών. Σας ευχαριστώ όλους και θα συνεχίσουμε στις 3.